δεν μπορούμε να τους περιμένουμε όλους. Είχαμε και μεγάλη συνεδρία σήμερα το πρωί με γεμάτη αίθουσα για τον αθλητισμό. Ελπίζω να ενδιαφέρουν εξίσου και τα άλλα ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει χαίρομαι για όσους έχουν έρθει, για τους λίγους που έχουν έρθει, που τουλάχιστον ενδιαφέρονται θα έχουμε την ε, ευκαιρία να έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Στην πρώτη σειρά δεν ακούγονται τα ακουστικά. Πρέπει να πάτε λίγο πίσω. Εντάξει, ναι, εμένα με καταλαβαίνεις, αλλά θα ακουστούν και γαλλικά και τέτοια διάφορα. Δεν ξέρω αν μας ακούει κανένας τεχνικός, μας ακούει, δεν μας ακούει. Να κάνουμε κάτι εδώ για τους ανθρώπους. Ε, γιατί δεν ακούγεται τίποτα στην πρώτη σειρά παρόλα αυτά. Ξεκινάμε. Χαιρόμαστε για το ότι είναι εδώ η Επιτροπή σα. Ε, και έχουμε βεβαίως και την Επίτροπο την υπεύθυνη για την ψηφιακή ατζέντα και τον πολιτισμό. Ζήτησε λοιπόν η Κομισιόν από τους ειδικού αυτούς να κάνουν κάποιες προτάσεις για το πώς θα μπορέσουμε να ασχοληθούμε καλύτερα με την ψηφιοποίηση, με το θέμα online και της διατήρησης της ε, πολιτικής μας κληρονομιάς, δηλαδή και με την Ευρωπαϊκή χαίρομαι για το ότι έχουμε τους τρεις σοφούς εδώ πέρα. Δεν είναι οι τρεις μάγοι με τα δώρα, είναι οι τρεις σοφοί από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ολλανδία Δηλαδή η κυρία Ελίζα Νίγκεμαν, Γενική Διευθύντρια της Γερμανικής Εθνικής Βιβλιοθήκης, ε, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Βιβλιοθηκών που διαχειρίζεται τη Γεροπεάνα, κατόπιν εδώ ο κύριος Μωρίς Λεβί από την Publis, μια γαλλική διαφημιστική εταιρεία. Publicis και μετά ο Ζακ Ντεντέκερ, συγγραφέας. Θεατρικός συγγραφέας. Δεν είναι εδώ. Εδώ είναι. Έρχεται. Έρχεται. Er Οπότε, οι τρεις σοφοί μόλις ολοκλήρωσαν μια διαβούλευση online και μετά στις 28 Οκτωβρίου είχαμε και την διαβούλευση και όπως ξέρετε τα θέματα τα οποία καλύφθηκαν εκεί συμπεριλαμβάναν την δυνατότητα της χρηματοδότησης, της ψηφιοποίησης, της ΣΔΙΤ και βεβαίως ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και αδειοδότησης. Και ομάδα προβληματισμού θα κάνει κάποιες προτάσεις στο τέλος του έτους και χαιρόμαστε που σήμερα θα ακούσουμε ήδη κάποια πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω τους τρεις σοφούς να μιλήσουν από 10 λεπτά και να μας πούν ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματά τους. Ξεκινάμε με, τον κύριο Μωρίς Λεβί. Έχετε τον λόγο. Ε, μπορείτε να μιλήσετε τη μητρική σας αν θέλετε. Θα μιλήσω γαλλικά. Σήμερα το πρωί μιλήσατε για κακά πνεύματα. Σήμερα θα μιλήσω για καλά πνεύματα με μια ένα πλεόνασμα κουλτούρας που το διακρίνει. Μετά από την πρόσκληση της κυρίας Κρούς και, του, και της κυρίας Βασιλείου, ξεκίνησαν οι εργασίες που αναφέρατε το Μάιο του ενεστώτος έτους και βρισκόμαστε στο τέλος της ε, εργασίας μας, του εγχειρήματος αυτό. Αν είμαστε σοφοί ή όχι δεν το ξέρω. Πάντως προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό και να το προσεγγίσουμε καταρχήν με κάποια αφέλεια και κατανοήσαμε στη συνέχεια ότι από πολλές πτυχές είναι ένα αχανές πρόβλημα. Υπάρχει και μια πάρα πολύ ισχυρή συγκινησιακή διάσταση γιατί πρόκειται, γιατί πρόκειται για την ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά και έχει να κάνει με τις βαθιές ρίζες και τη ζωή των Ευρωπαίων. Δεν ξέρω αν είμαι σε θέση να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας σήμερα το απόγευμα, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχουμε την ευκαιρία να είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ώστε να σας παρουσιάσουμε την κατάσταση πραγμάτων, την κατάσταση προόδου των εργασιών μας. Η εντολή μας ήταν πραγματικά ευρύτατη, κάλυπτε πάρα πολλές πτυχές του προβλήματος, ουσιαστικά θέματα που έχουν να κάνουν με την χρηματοδότηση της της ψηφιοποίησης με το να υπάρξει ένα μέλλον στα πολιτιστικά αυτά θέματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επίσης επρόκειτο για να μπορέσουμε να καθορίσουμε τις ε, προϋποθέσεις και τις συνθήκες μιας εταιρικής σχέσης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και να αποσαφηνίσουμε το πώς θα μπορούσαμε να μεταφέρουμε στον ψηφιακό κόσμο και έργα τα οποία είναι ε, προστατεύονται από copyright και αυτά τα οποία είναι όπως λέμε ορφανά διότι έχει εκπνεύσει το copyright τους. Επομένως να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την προσβασιμότητα διαφόρων έργων στο διαδίκτυο και όχι αποκλειστικά και μόνο πτυχές οι οποίες συνάπτονται με την προσέγγιση μιας συγκεκριμένης χώρας. Ξεκίνησαμε λοιπόν το Μάιο όπως σας είπα εργαστήκαμε σε βάθος, πραγματικά σε βάθος και αυτό το οποίο ανακαλύψαμε με κάποιες ανησυχίες παράλληλα είναι ότι τόσο το, η πολιτιστική διάσταση όσο και η οικονομική διάσταση του προβλήματος είναι τεράστιες. Και είτε σκεφτόμαστε υπομορφή αριθμητικών στοιχείων είτε σκεφτόμαστε σε επίπεδο προκλήσεων για την κουλτούρα μας είναι πράγματι αχανεστό πρόβλημα. Ένα δεύτερο στοιχείο. Ενώ εμείς είχαμε αποδεχθεί σε αυτή την εργασία υπήρξαν και άλλοι οι οποίοι προχωρούν με μεγάλα και γοργά βήματα. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε σε αρκετά ταχείς δράσεις <clears throat> και δεν είναι ούτε απλό ούτε προφανές το πώς θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Πώς αντιμετωπίσαμε λοιπόν το εγχείρημα αυτό την αποστολή μας. Καταρχήν με απόλυτα ανοιχτό πνεύμα, χωρίς απριόρι, χωρίς προκαταλήψεις, ανεξάρτητα από τα προβλήματα τα οποία μπορούν να τεθούν σε σχέση με τους εμπλεκόμενους στον χώρο αυτό το πολιτιστικό, ανεξάρτητα από τη χώρη προέλευσης αυτού του φορέα, εμείς δεν έχουμε καμία προκατάληψη απέναντί του, όπως δεν έχουμε και καμία προκατάληψη έναντι των εκδοτών, των καλλιτεχνικών δημιουργών. Ξεκινήσαμε όλοι με την ιδέα μιας μεγάλης φιλοδοξίας και με στόχο να δούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσαμε να δώσουμε απαντήσεις στα πολλαπλά προβλήματα, λαμβάνοντας υπόψη και την ε, εφαρμοσιμότητα που έχουν σε όλους τους φορείς του τομέα αυτό και επίσης να αναζητήσουμε αρχές οι οποίες θα είναι σχετικά απλές και εύληπτες και συγχρόνως θα οδηγούν σε λύσεις οι οποίες είναι εφικτού χαρακτήρα. Μεταξύ μας λοιπόν καθορίσαμε μια προσέγγιση η οποία είναι και οραματιστική και πραγματιστική. Θέλαμε να είμαστε οραματιστές γιατί ο κόσμος αλλάζει. Είναι ένας κόσμος ο οποίος είναι ρευστό, αλλάζει συνέχεια. Συγχρόνως όμως πραγματιστητές γιατί υπάρχουν και στοιχεία της πραγματικότητας που δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε και να απαραίτητο να λάβουμε υπόψη μας. Ως εκ τούτου, <clears throat> προετοιμάσαμε μια σειρά από οι οποίε κινούνται προ την κατεύθυνση του οραματισμού πραγματισμού, είναι ισχυρέ και σε επίπεδο αρχών, αλλά λαμβάνουν υπόψη συγχρόνω και την πραγματικότητα. Σήμερα δεν είμαστε σε θέση να σα πούμε ποιε ακριβώ θα είναι αυτέ οι συστάσει, αλλά είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε στα ερωτήματά σα. Τι ακριβώ έχουμε κάνει. Προβήκαμε σε μία διαβούλευση η οποία θέλησαμε να είναι όσο δυνατόν πιο πλούσια, πιο πλήρης θέλαμε να προσελκύσουμε αυτούς που πραγματικά ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό χώρο και όχι τους περίεργους. Θέλαμε να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι οποίοι θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διαβούλευση ήταν αυτοί οι οποίοι είχαν να πούνε κάτι ενδιαφέρον και ήταν έτοιμοι να συμπληρώσουν όλο το ερωτηματολόγιο που τους υποβάλαμε. Μια πρώτη έκπληξη ήταν τα πρότυπα της Κομισιόν για τον αριθμό των συμμετεχόντων 1228 για την ακρίβεια αλλά μέσα σε αυτούς δεν υπήρχαν οι παραδοσιακές ομάδες πιέσεων και χαιρόμαστε για τις πληροφορίες που μας έδωσαν αυτοί οι άγνοι λομπίστες, αλλά επίσης υπήρχαν και Ευρωπαίοι πολίτες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι μας προσέθεσαν και τις δικές τους μέρινες και ανησυχίες. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο θέλω να τονίσω, κυρία Πρόεδρε, είναι ότι διοργανώθηκε μια δημόσια κρόαση η οποία διαδόθηκε στο διαδίκτυο με 100 περίπου συμμετέχοντες που ήταν μια σημαντική στιγμή για την ομάδα εργασία μας γιατί είδαμε κάτι το ιδιαίτερα έντονο να υπάρχουν οι ηγέτες στον επαγγελματικό αυτό τομέα που μας διεφώτισαν τα μάλα. Δεν μετανιώνουμε καθόλου λοιπόν για αυτή την ακρόαση, ήταν μια ακρόαση άκρος ενδιαφέρουσα. Επίσης, ήρθαμε σε επαφή με τους αρμόδιους υπουργούς των κρατών μελών οι οποίοι <clears throat> συνεπλήρωσαν τον κατάλογο των ετοιμάτων που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και οι οποίοι μας πρόσθεσαν και τα δικά τους, μας έδωσαν και τα δικά τους φώτα σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία έχουν τη μεγαλύτερη σημασία σε εθνικό επίπεδο για καθένα από αυτούς. Τι μπορούμε να πούμε λοιπόν από, όλα αυτά τώρα. Η πρώτη παρατήρηση που θέλω να κάνω είναι ότι αρχίσουμε να έχουμε κάποιες ενδείξεις για τα αριθμητικά ποσά. Ζητήσαμε να υπάρχει μια μελέτη που έγινε από μια αγγλική εταιρεία που θα μας δώσει τα οριστικά της αποτελέσματα σε μερικές μέρες. Αλλά θα αρχίσουμε να έχουμε σύντομα αριθμητικά στοιχεία τα οποία θα κάνουν μέσα εισαγωγικά να χλιμιντρήσουν όλοι βλέποντας πόσα είναι τα οικονομικά διακυβευόμενα. Επίσης, βλέπουμε την τεράστια λιτότητα μέσα στην οποία βρίσκονται τα κράτη-μέλη για να μην πούμε την αδιοτσεπία των κρατών μελών και το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δημόσια κονδύλια για τον τομέα αυτό υπάρχει πραγματικά μια πρόκληση που θα είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσουμε σε σχέση με την χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης των πνευματικών έργων. Και παράλληλα θα τεθούν σημαντικά θέματα και ερωτήματα για το πώς θα χαράξουμε την οριοθετική γραμμή και πού θα τρέχει ο δρομεύς σε σχέση με την ε, εταιρική σχέση δημοσίου ιδιωτικού τομέα, ώστε να βρισκόμαστε σε μια οδική, οδηγό που επιτρέπει τον έλεγχο από τους Ευρωπαίους και τους πολιτιστικούς φορείς του πολιτιστικού περιεχομένου και την πρόσβαση από ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο ακροατήριο, ενώ συγχρόνως θα είμαστε δίνον ε, κίνητρα στους, ε, δημόσιους, στους ιδιωτικούς φορείς ώστε να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν αυτό το εγχείρημα. Εμείς συνειδητοποιούμε ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Περαιτέρω, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το θέμα του copyright, των συγγραφικών δικαιωμάτων και ιδίως αυτού το οποίο εγώ ονομάζω της μαύρης τρύπας του 20ου αιώνα. Με ποιο τρόπο λοιπόν θα προσπαθήσουμε, θα μπορέσουμε να ψηφιοποιήσουμε όλο αυτό το περιεχόμενο και πώς θα εξασφαλίσουμε ότι αυτό το περιεχόμενο θα είναι προσβάσιμο σε όλους με σεβασμό των πνευματικών δικαιωμάτων των πνευματικών δημιουργών και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο εμεί έχουμε προχωρήσει, έχουμε συγκεκριμένες ιδέες και σε σχέση με το οποίο θα έχουμε σαφείς συστάσεις να διατυπώσουμε. Υπάρχει περαιτέρω μια άλλη πτυχή που αφορά τα έργα τα οποία δεν βρίσκονται στην αγορά, τα λεγόμενα ορφανά έργα για τα οποία η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη. Διότι ποικίλει η σχετική νομοθεσία από κράτο μέλο σε κράτο μέλο σε σχέση με αυτά τα ορφανά έργα. Τέλο, υπάρχει ακόμα μια ουσιώδη πτυχή του προβλήματο, την οποία επίση δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε. Ότι δηλαδή όταν ψάβομαι τον ψηφιακό χώρο, έχουμε μπροστά μας ένα χώρο ο οποίος είναι ρευστός, κινητικός, πρωτεϊκός και ο οποίος αλλάζει με επιτάχυνση πολύ υψηλή. Ως εκ τούτου μπορεί να καταλήξουμε να κάνουμε σημαντικές επενδύσεις οι οποίες πολύ γρήγορα θα είναι πε... πεπαλαιωμένες. Επομένως, το θέμα της ταχείας ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και το θέμα της ταχείας υλοποίηση αυτών των ψηφιακών εργασιών. Αυτό είναι από τα θέματα για τα οποία εργαζόμαστε. Εν πάση περιπτώσει, η Ευρωπαϊάνα μα απασχόλησε πάρα πολύ. Η Ευρωπαϊάνα είναι μια ιστοσελίδα όπου μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε βιβλία σε ένα επίπεδο το οποίο είναι κοντά στο επίπεδο του Google. Δυστυχώς δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο του Google. Ξέρουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά, πάντως η Ευρωπαίανα δίνει πρόσφαση σε 1.200.000 βιβλία, ενώ το Google δίνει μονάχα σε 1.500. Δεν απέχουμε λοιπόν πολύ από το Google, αλλά δεν πρέπει να δει το θέμα κανείς μονάχα από αριθμητική πλευρά. Βρισκόμαστε στην τελική φάση των εργασιών μας θα κάνουμε ακόμα μερικές συνεδριάσεις, η επόμενη την επόμενη εβδομάδα. Εργαζόμαστε μαζί με τον Ζακ και την Ελισαμπέτ Νιγκεμάν και πιστεύω θα είμαστε σε θέση να έχουμε περατώσει την εκθέσή μας λίγο πριν από τα Χριστούγεννα με την θέληση ότι με την πρόθεση να μπορείτε να τη διαβάσετε προσεκτικά τις ημέρες των διακοπών ή τις βροχερές ημέρες ώστε και με τα σχόλιά σας και εμείς να μπορέσουμε να την φέρουμε σε μια Οπότε η κυρία Αντρούλα Βασιλείου, η οποία είναι ο εντολοδόχος κατά κάποιο τρόπο αυτής της εργασίας, θα έχει το τελικό έγγραφο στις αρχές του Ιανουαρίου. Θα θέλαμε να έχουμε και περισσότερο χρόνο για την περάτωση αυτής της εργασίας αλλά θεωρούμε ότι με αυτά τα οποία κάνουμε θα δημιουργήσουμε το υπόβαθρο το οποίο θα επιτρέψει να φωτιστεί λίγο καλύτερα αυτό το τόσο αχανές θέμα. Δίνω το λόγο στην Ελίζαμπεθ και στον Ζακ για να μπορέσουν να συμπληρώσουν αυτά τα οποία είπα. Ευχαριστώ κύριε Λεβί μου. Ähm, κύριε Νίγκερμαν, ευχαριστώ. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα Απλά ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ευκαιρία που μας δίνετε και ευχαριστώ να απαντήσουμε σε ερωτήσεις και ρεθίσματα για την περαιτέρω εργασία μας. Ωραία. Τώρα χαιρετίζω και τον συγγραφέα. Έχετε τον λόγο και μιλήστε βεβαίως ε, περισσότερο εφόσον και η κυρία δεν θα μιλήσει. Νομίζω ότι όλα ε, εξετέθησαν από τον πρόεδρό μας Η εμπειρία αυτή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, αλλά είναι και στο ύψος των προσδοκιών μας. Το θέμα αυτό τέθηκε μόνο του θα έλεγα και έτσι η επιτάχυνση της ενασόλησής μας με το συγκεκριμένο θέμα είναι κάτι το οποίο ε, έχετε υπόψη σας πλέον, να προσπαθήσετε να σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και νομίζω ότι ο προηγούμενος ομιλητής το εξήγησε πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε τότε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με όλους τους συναδέλφους, τους ευρωβουλευτές. Ε, λέω και πάλι στους συναδέλφους εδώ μπροστά δεν δουλεύουν τα ακουστικά. Άμα θέλετε καθίστε λίγο πιο πίσω. Η κυρία Τρούπελ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Δόρης και θέλω να ευχαριστήσω και τους εμπειρογνώμονές μας. Ευχαριστώ την Επιτροπή των Σοφών. Κύριε Λεβί, έχετε παρουσιάσει τις τεράστιες προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιόν μας. Ο στόχος μας ήταν ακριβώς να επιφορτήσουμε την Επιτροπή των Σοφών ώστε να μας δώσουν όχι μόνο το μέγεθος των προκλήσεων, αλλά να μας δώσουν και δρόμους για να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα πολύπλοκα προβλήματα που έχουμε μαζί μας. Ξέρω ότι δεν έχετε τελειώσει ακόμα την εργασία σας, αλλά νομίζω ότι έχετε διεξέλθει όλα τα μεγάλα ερωτήματα και τις μεγάλες προκλήσεις. Γι' αυτό μπορώ να διατυπώσω κάποια ερωτήματα με την ελπίδα ότι θα μου δώσετε κάποιες έστω προσωρινές απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Ένα μέρος της πολιτικής συζήτησης για τα θέματα αυτά περιστρέφεται γύρω από το εξή σημείο. Όταν θέλει κανείς να εξασφαλίσει τη δημόσια πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή, επομένω το συνολικό όγκο της Ευρωπαϊκής Πολιτιστική Κληρονομιάς, τίθεται το θέμα της χρηματοδότησης, αλλά και το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, που έχουμε ένα διαφορετικό σύστημα από τις Ηνωμένες Πολιτείες που υπάρχει το μοντέλο copyright αλλά και fair use, δικαιώματα χρήσεως. Έχουμε διαφορετικές ε, παραδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πνευματικών δημιουργών. Επομένως, από τον πολιτικό χώρο υπάρχει μια ε, αίτηση από την πολιτική πλευρά να υπάρξει η, η ευρύτερη δυνατή αντιμετώπιση των προβλήματων των πνευματικών δικαιωμάτων ώστε η ψηφιοποίηση να καλύψει ως το δυνατόν και περισσότερα έργα. Βέβαια, το τωρινό σύστημα δεν είναι επαρκές. Θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά, να υπάρξουν συστήματα αμοιβαία αναγνώρισης μεταξύ ε, κρατών μελών, τρόποι με τους οποίους θα, θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Ξέρω τώρα ότι από εσά μπορεί να προκύψει κάποια λύση στα πλαίσια της εργασίας σας. Και έρχομαι και πάλι σε ένα θέμα το οποίο πάντα παράγει κάποιες αντιφάσεις όταν ακούμε διάφορε απόψει. Και εγώ θα ήθελα να ξέρω αν εσεί ω τρει σοφοί έχετε να προβλέψετε, να προτείνετε μάλλον, μία πρόταση ή αν έχετε κάποιες ε, κατά κάποιο τρόπο κατευθύνσεις στις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε ώστε όλη αυτή η συζήτηση να γίνει λίγο πιο απτή και συγκεκριμένη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους ομιλητές και την Πρόεδρο. Εντάξει. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Έχω μια ερώτηση μετά από αυτό το οποίο είπε η κυρία Τρούπελ γιατί τα πνευματικά δικαιώματα μας απασχολούν με πολλούς τρόπους και η Ευρώπη είναι μία από τις πιο πολυπίκυλες πολιτισμικά περιοχές κάτι το οποίο νομίζω δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως την παγκόσμια οικονομία και αυτό σχετίζεται με το ότι η ψηφιακή αγορά της Ευρώπης δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις εντός και εκτός της Ευρώπης. Και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζητάμε συχνά την αυστηρότερη τήρηση των υφισταμένων νόμων, ενώ υπάρχουν άλλες φωνές που ζητούν μεταρρύθμιση και βέβαια αυτό σχετίζεται με την παλέτα επιλογών που ανέφερε η κυρία Τρούπελ για την ανταμοιβή των καλλιτεχνών. Οπότε αναρωτιόμουν τι μεταρρυθμίσεις έχετε συναντήσει και τι έχετε μάθει από τους καλλιτέχνες. Γιατί ακούμε τους λομπίστες που λένε πως εκπροσωπούν τους καλλιτέχνες αλλά δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθες. Και όταν κοιτάτε τα νούμερα και τους προϋπολογισμούς ε, περί ψηφιοποίησης, εάν λαμβάνετε υπόψη το κόστος ευκαιρίας, ε, δηλαδή τι θα γίνει αν ε, δεν εναρμονίσουμε την αγορά αυτή στην Ευρώπη και πώς θα περάσουμε από 27 διαφορετικά νομικά συστήματα σε ένα ευρωπαϊκό και τις δυσκολίες που σχετίζονται με αυτό κατόπιν εάν έχετε διδαχθεί από βέλτιστες πρακτικές και την έννοια βεβαίως της εύλογης χρήσης όπως ισχύει στο Αμερικάνικο Δίκαιο Πνευματικής Διοκτησίας ο Πόλωνος συναλφός μας, ο κύριος Μπόρης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω λοιπόν τους τρεις εμπειρογνώμονες για την παρουσίασή τους. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα για την πολιτιστική κληρονομιά. Κάτι το οποίο δεν αφορά μόνο την λογοτεχνία, αλλά και, την, ε, και τις οικαστικές τέχνες η Ευρωπαϊκή είναι ένα τμήμα του ευρύτερου πάζολ, αλλά το θέμα είναι να υπάρξει δυνατότητα πρόσβασης και στα έργα τέχνης γενικότερα. Οικαστικά, χάρτες, οπτικοακουστικά, ντοκιμαντέρ, κινηματογράφος, τα πάντα μπορούμε να βρούμε στο διαδίκτυο. Έρχεται λοιπόν η ερώτησή μου εδώ η οποία ταιριάζει με την ερώτηση της κυρίας Τρούπελ. Τι είδους επιχειρηματικό πρότυπο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε, να προκρίνουμε σε σχέση με το σεβασμό ε, της πνευματικής ιδιοκτησίας και σε σχέση με την ψηφιακή ευρωπαϊκή ατζέντα. πώς θα μπορέσετε να ενσωματώσετε τα οπτικοακουστικά υλικά σαν παράδειγμα και άλλες μορφές ευρωπαϊκής τέχνης και να τα συνδυάσετε με τα επιχειρηματικά πρότυπα. Λοιπόν, θα κάνω και εγώ μια ερώτηση και μετά θα τελειώσουμε. Θα ήθελα να γνωρίζω, είπατε ότι είχατε έρθει σε επαφή και με τους υπουργούς το απόγευμα της ακρόασή σας. Τι είπαν οι υπουργοί. Είναι έτοιμοι να σας δώσουν πρόσβαση στο πολιτιστικό κληροδότημα της Γερμανίας, της Γαλλίας. Εγώ έχω αμφιβολίες. Θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό είναι έτοιμοι να ανοίξουν τους εθνικούς τους θησαυρού και αν υπάρχει κάτι το οποίο θα τους τροχοπεδίσει σε αυτή την κατεύθυνση. Σε ποιο θα δώσω τώρα το λόγο. Α, κύριε Λεβί, παρακαλώ με την ε, άδειά σα θα απαντήσω σε ορισμένα στοιχεία των ερωτήσεών σα, και μετά θα ήταν πρέπον και ορθό η Ελισάβετ Νίκεμα να σα δώσει περισσότερε πληροφορίε. Δεν μπορώ να σας πω εγώ αυτά τα οποία μπορούν να κάνουν οι Υπουργοί. Η συζήτηση είχε συγκεντρωθεί κυρίως στο τι περιμένουν από μας και στις ερωτήσεις τις οποίες μας έθεσαν και τα θέματα τα οποία θα ήθελα να συμπληρώσουμε στις εργασίες μας. Η αίσθηση η οποία μου δημιουργήθηκε είναι ότι καταρχάς υπήρξε μια εκπληκτική από πλευρά τους εμπλοκή και ενδιαφέρον. Όλοι πήραν μέρος στη συζήτηση με πολύ δραστήριο τρόπο και αυτό το οποίο διαπίστωσα επίσης είναι ότι ορισμένοι είχαν ζητήσει το λόγο για να παρέμβουν και στο τέλος μίλησαν πολύ περισσότεροι. Ήταν εντός θέματος και το θέμα δεν ήταν καθόλου ελαφρύ και εύκολο. Μου έδειξαν λοιπόν ότι υπολογίζουν τα θέματα αυτά με πολύ σοβαρό τρόπο. Δεύτερη παρατήρηση. Διάβασα την έκθεση της κυρίας Τρούπελ όπως και η διπλανή μου. Μας δόθηκε η έκθεση αυτή μαζί με άλλα σημαντικά στοιχεία στα οποία και έγγραφα στα οποία είχαμε πρόσβαση και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν σαν καύσιμο θα έλεγα για τη δική μας μελέτη. Το θέμα των συγγενικών δικαιωμάτων είναι ένα θέμα ιδιαίτερα περίπλοκο Καλό θα είναι ο Ζακ να πάρει το λόγο πάνω σε αυτό. Γιατί όχι μόνο υπάρχουν κάποια θέματα που διαφέρουν σε κάθε χώρα από τις άλλες, αλλά τίθεται και ένα ευρύτερο θέμα για την καλλιτεχνική δημιουργία στο μέλλον, την οποία δεν θα πρέπει να αποθαρρύνουμε. Το τρίτο σημείο, το οποίο σύντομα θα θέσω, είναι αυτό το οποίο έθεσε η κυρία Σάκη αν άκουσα καλά και αφορά την, το επιχειρηματικό μέλλον και τις εμπορικές δυνατότητες. Το θέμα αυτό του οικονομικού εμπορικού δυναμικού το θίξαμε κατά τη διάρκεια του, του γεύματος και πιστεύουμε ότι υπάρχουν αρκετά σημαντικά θέματα τα οποία μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας σαν δυνατότητα απόσβεσης επενδύσεων εφόσον είμαστε σε θέση να κινητοποιήσουμε το επιχειρηματικό πνεύμα των Ευρωπαίων. Και το θέμα του κύριου Μπάρις για το ε, οπτικοακουστικό περιεχόμενο είναι κάτι το οποίο τέθηκε επίμονα από πολλούς από τους υπουργούς κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος. Νομίζω ότι πραγματικά σοφοί παρακαθήμενοι μου να πάρουν το λόγο. Η είναι κασοφός τώρα. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα περισσότερο για τα οπτικοακουστικά. Η αίσθηση πως η Ευρωπαϊκή παραδείγματο χάρη δεν είναι αρμόδια και υπεύθυνη γι' αυτό, προέρχεται από το ότι όλα τα οπτικοακουστικά έργα δημιουργήθηκαν τον 20ο αιώνα. Δηλαδή η τεχνολογία δεν υπήρχε για να διατηρηθούν αυτά στο αρχείο και αυτό ακριβώς είναι το μεγάλο θέμα, το θέμα των δικαιωμάτων του δημιουργού Γι' αυτό ακριβώς υπάρχει μεγάλος αριθμός έργων ε, για τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεκαθαρίσουμε όλους τους δικαιούχους των δικαιωμάτων και να τους βρούμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για το πόσο σημαντικά είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή αφενός η ανάγνωση του περιεχομένου και αφετέρου το να ξεκαθαρίσουμε τα δικαιώματα. Το πιο ακαθόδες νομίζω είναι και είναι δυσκολότερο νομίζω αυτό από το οικονομικό είναι τα δικαιώματα και τι θα κάνουμε με τυχόν ε, έργα τα οποία δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Και θα ήθελα εδώ πέρα να δώσω τον λόγο στον ε, κύριο Ντεντέκερ. Ευχαριστώ Ελισάβετ. Προσπαθούμε να αναλύσουμε τις διαφορετικές προβληματικές που εκθέτει το συγκεκριμένο θέμα. Είναι διαφορετικές μεταξύ τους, ποικίλουν, είναι περίπλοκες όπως είπε ο Μωρίς Λευδή και είναι ταυτόχρονα και ιδιαίτερα πρόσφατες. Νομίζω ότι σε αυτήν εδώ την συνάντηση δεν θα συμβαίνει πολύ συχνά τα θέματα αυτά να τίθενται με τέτοια οξύτητα. Αυτό οφείλεται και στην τεχνολογική διάσταση που μας οδηγούν να αντιμετωπίζουμε κατά μέτωπο θέματα που κρύβαμε συστηματικά στο παρελθόν όπως το θέμα των συστημάτων συλλογής ε, των ε, πνευματικών δικαιωμάτων. Υπάρχουν διαφορετικές ρυθμίσεις, διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις Μέσω του διαδικτύου και μέσω της κατάργησης των συνόρων δεν μπορούμε να αρκεστούμε πλέον με την συγκατοίκηση διαφορετικών συστημάτων σε ένα συγκεκριμένο εδαφικό χώρο. Η ώρα της αλήθειας έφτασε πλέον. Το θέμα τίθεται σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων της Ένωσης και στο δικό σας. Εμείς δεν είμαστε παρά πολύ απλοί συνεισφορείς, πληροφοριοδότες σε εισαγωγικά στην ουσία εμείς αντιμετωπίζουμε ε, ε, ε, την προβληματική αυτή σε καθημερινή βάση στις δραστηριότητες τις οποίες έχουμε ο καθένας. Αλλά εσείς και στο Συμβούλιο Υπουργών ασχολείστε με τα θέματα αυτά και θα πάρετε αποφάσεις. Ο Μωρίς Λεβί εξήγησε ότι αυτό το Συμβούλιο Υπουργών μας άφησε μια εξαιρετική εντύπωση ότι αυτοί που ήταν εκεί δεν είχαν έλθει απλά για το μεσημεριανό φαγητό αλλά είχαν πράγματι ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα θέματα σε βάθος και πήραν το λόγο και ε, ήταν περίπλοκες και λεπτομερείς ε, οι παρεμβάσεις τους αντίστοιχες με αυτά που ακούσαμε εδώ. Το θέμα αυτό ε, απασχολεί πολύ κόσμο. Θα πρέπει πάντως το θέμα να μπει και σε τέτοιου είδους αίθουσες συνεδριάσεων η Επιτροπή Πολιτισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να δείξει και να αποδείξει ότι είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Και γι' αυτό είναι μια ευκαιρία κυρίως για σας και όχι τόσο για μας να μπορέσετε να πάρετε αποφάσεις γύρω από τα θέματα αυτά. Θα κάνετε πολλές συζητήσεις, θα ακούσετε αντιφάσεις ε, θα υπάρξουν αντιτιθέμενες φιλοσοφίες σχετικά με τον ορισμό των συγγενικών ή πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα και θα δούμε στο τέλος πώς θα καταλήξουμε. Ακούσουμε και άλλη μια ερώτηση από την κυρία Τρούπελ. Ναι, είπατε πάλι πως όλα αυτά την κυρια τριπελ ναι μεγάλες συγκρούσεις και ε, θα έχουμε συναρπαστικές συζητήσεις. Εδώ για ένα μισή χρόνο ασχολούμαστε με αυτό το θέμα. Εγώ περίμενα από εσά να μας πείτε τουλάχιστον κάποια σενάρια ή επιλογές. Για να μπορέσουμε να σκεφτούμε με βάση κάποια κείμενα το προς τα που θα πάει αυτή η υπόθεση. Δηλαδή το βασικό ερώτημα θα πρέπει ε, να είναι να κάνουμε για αυτά τα ορφανά έργα μια γενική εξαίρεση ή να κάνουμε μια αναζήτηση για να αποζημιωθούν αναλόγως οι δημιουργοί. Γιατί άλλοι λένε πρέπει να κάνουμε μια γενική εξαίρεση και μετά υπάρχει τεράστιο οικονομικό όφελος και από την άλλη υπάρχουν αυτοί που λένε πως δεν μπορούμε εδώ πέρα να ξεχάσουμε την έννοια της πνευματικής ιδιοκτησίας, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω μετά τις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που κάνατε εσείς να μας παρουσιάσετε τουλάχιστον κάποιες επιλογές για να μπορέσουμε να συζητήσουμε. Είναι μεγάλη πρόκληση. Ότι είναι πρόβλημα το ξέραμε και από μόνοι μας, να σας πω την αλήθεια. Ευχαριστώ. Βεβαίω αλήθεια είναι πως δεν έχουν ολοκληρώσει τις συζητήσεις του οι τρεις σοφοί. Ελπίζω λοιπόν να μπορέσετε να βρείτε ένα σημείο ε, ισορροπίας. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν είμαι και νομικός. Σας ζητάμε τον τετραγωνισμό του κύκλου. Όταν μιλάμε με συγγραφείς ε, ακούω να μου λένε από τη μία δεν έχει καμία σημασία το copyright, το θέλω το βρίσκω εγώ στο ίντερνετ και είμαι σίγουρος πως υπάρχουν άνθρωποι που το θεωρούν πάρα πολύ καλό. Εγώ το βρίσκω τρομερό. Αλλά βεβαίω αν θέλει κάποιο να γίνει γνωστό είναι η καλύτερη πλατφόρμα. Αλλά αν θέλει να βγάλει και λεφτά ε, είναι τελείω διαφορετικά τα πράγματα. Οπότε εγώ το βρίσκω δύσκολο. Γι' αυτό ζητήσαμε από εσά του τρει ε, σοφού να βρείτε ποιο είναι ο σωστό ο δρόμο. Όπω έκαναν οι τρει μάγοι από τη Διθλεέμ. Ελπίζω. Εντάξει, δεν είπα να κάνετε θαύματα, το αντιλαμβάνομαι αυτό. Ελπίζω λοιπόν εκεί που θα πάτε διακοπέ το χιόνι, τα Χριστούγεννα, να βρείτε κάποια σοφία έτσι ώστε Ιανουάριο, Φεβρουάριο να μπορέσετε να μας χαράξετε ένα δρόμο γιατί θα αποτελέσετε βάση και για τον κύριο Μπαρνιέ, όχι μόνο για την κυρία Βασιλείου, γιατί και αυτός πρέπει να υποβάλει μια οδηγία για το copyright, η οποία πρέπει βέβαια να ανταποκρίνεται στις απαιτήσει μας. Δεν θα μιλήσω παραπέρα. Χέλγα, δεν πήρες απάντηση. Νομίζω ε, δεν ήθελες κιόλα. Δεν θέλουμε σήμερα απάντηση. Ελπίζω να σας έρθει έτσι η θεία. Φώτιση τις ερχόμενες εβδομάδες και να έχουμε μια απάντηση ε, του χρόνου. Σας ευχαριστώ που αναλάβατε λοιπόν αυτό το καθήκον και Είμαι σίγουρος ότι θα οδηγηθούμε σε ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Ε, τέλειο όχι, δεν μπορεί να ικανοποιηθούν όλοι. Έτσι είναι αυτά στην πολιτική. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank και merci Και, και τώρα με μεγάλη χαρά μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. Αν έχετε κι άλλες ε, υποχρεώσεις ε, δεν θα σας ε, κακολογήσει κανείς. Έχουμε στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης και χαίρομαι πάρα πολύ που η αντιπρόεδρος του, της Κομισιόν, η κυρία Κρούς, είναι μαζί μας. Έχουμε ήδη συζητήσει μαζί της στο παρελθόν, κατ' επανάληψη. Θα της δώσω αμέσως το λόγο. Γνωρίζει τα θέματα τα οποία μας απασχολούν. Ξέρει ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και μπορεί να μας πει ποια είναι τα εγχειρήματα που θέλει να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα της ψηφιακής, ε, του ψηφιακού θεματολογίου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ντόρις. Αγαπητά μέλη της Επιτροπής Πολιτισμού, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα όλα τα μέλη της Επιτροπής και όλους αυτούς οι οποίοι ενδιαφέρονται στον τομέα αυτό των πολιτιστικών θεμάτων και ιδιαίτερα για τις δραστηριότητες μας που έχουν να κάνουν με το ψηφιακό θεματολόγιο. Δεν κομίζω ψηφιακή γλάφκα σε εσά. Αν σας πω ότι γνωρίζω ότι ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για τις πρωτοβουλίες σας, όλα αυτά τα θέματα που εμπίπτουν στο δικό μου χαρτοφυλάκιο και επίσης είχα την ευκαιρία να έχω και διμερείς ε, ε, συζητήσεις με πολλούς για το σύστημα εκπομπών μέσα στα πλαίσια της ψηφιακής ατζέντα και τα θέματα του, των ραδιοσυχνοτήτων ψηφιακού χαρακτήρα. Τον Ιούνιο είχαμε επίση την, ευκαιρία, την ευκαιρία να παρουσιάσω το ψηφιακό θεμετολόγιο. Ξέρετε όλοι ότι είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Εν πάση περιπτώσει αυτός ο στόχος μας, μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη και να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε μέσα στα πλαίσια του εγχειρήματος της Ευρώπης 2020. Πρέπει να παίξει κάποιο ρόλο σε αυτά και το ψηφιακό θεματολόγιο. Θέλω να μιλήσω σε σας σήμερα για τα πρώτα μέσα, τα πρώτα μέτρα μάλλον καλύτερα, εφαρμογής του ψηφιακού θεματολογίου. Μιλάω για τις ευρυζωνικές ε, επικοινωνίες και το πρόγραμμα για τις ραδιοσυχνότητες και επίσης θέλω να ανταλλάξω και πληροφορίες μαζί σας για το πρόγραμμα που έχουμε για την ψηφιακή ατζέντα για τον επόμενο χρόνο το 2011 όλοι συμφωνήσαμε ότι η οικουμενική ευρυζωνική πρόσβαση στο ίντερνετ θα παίξει μεγάλο ρόλο, δημιουργώντας μια πλατφόρμα που υποστηρίζει την καινοτομία σε όλη την οικονομία μας και μειώνοντας το ψηφιακό χάσμα. Έχω απόλυτη επίγνωση του γεγονότος ότι είναι πολύ περισσότερα τα διακυβευόμενα, δεν είναι μονάχα το θέμα της οικονομικής δραστηριότητας και δεν μπορούμε και όχι μονάχα της μείωσης του ψηφιακού χάσματος, αλλά Μιλάμε και για τις ανάγκες 500 εκατομμυρίων ανθρώπων στην Ευρώπη και πώς μπορούν να αποκτήσουν πληροφορία και πολιτιστικά αγαθά. Η ευρυζωνική επικοινωνία λοιπόν είναι ένα κομμάτι ενός καλαθιού από προτάσεις που έχει υποβάλει η Επιτροπή και μία είναι η σύσταση για, τις, ε, για την πρόσβαση νέα ε, νέας γενιάς και το άλλο είναι η πολιτική για τις ραδιοσυχνότητες στις επικοινωνίες. Η ανακοίνωση της Κομισιόν αναγνωρίζει ότι θα χρειαστούν σημαντικές επενδύσεις για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε υποδομή για ταχεία πρόσβαση στο ίντερνετ σε όλη την Ευρώπη. Χρειάζομαι προφανώς την υποστήριξή σας γιατί αυτό ήταν μια διακινδύνευση από την πλευρά της ε, Κομισιόν να εκδώσει μια τέτοια ανακοίνωση που τονίζει την ανάγκη των ευρυζωνικών επικοινωνιών, γιατί αν αυτέ δεν ευδοκιμήσουν, τότε θα έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η ανακοίνωση αυτή θεσπίζει ένα πλαίσιο για όλου του εμπλεκομένου και ενδιαφερομένου, είτε είναι τα κράτη-μέλη, είτε είναι ο ιδιωτικό τομέα, τοπικέ και περιφερειακέ αρχέ. Όλοι αυτοί οι φορεί θα πρέπει να συνεργαστούν από κοινού και εμεί μαζί του για να μπορέσουμε να επιτύχουμε του στόχου αυτού που έχουμε καθορίσει στην ανακοίνωση τη Κομισιόν. Στο ψηφιακό αυτό θεματολόγιο και που περιλαμβάνουν τις δεσμεύσεις μας. Θέλουμε φυσικά να συνεργαστούμε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Επίσης, τα, οι εθνικές, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να ε, δημιουργήσουν, να διαμορφώσουν εθνικά σχέδια για τις ευρυζωνικές επικοινωνίες. Επίσης, το κόστος των επενδύσεων σε ευρυζωνικές επικοινωνίες θα πρέπει να μειωθεί, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι δεδομένο το τωρινό κόστος, αν είμαστε επιτυχεί και αν και τα κράτη-μέλη είναι επιτυχή, θα πρέπει να υπάρξει κατάλληλο σχεδιασμό και συντονισμό σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για την βελτίωση των υποδομών, γιατί όλα αυτά θα βελτιώσουν τα μάλλα την κατάσταση. Ένα τρίτο στοιχείο είναι η χρήση του Περιφερειακού Ταμείου, του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Ανάπτυξη τη Υπέθρου για την ε, δημιουργία υποδομών. Και αυτό είναι κάτι το οποίο επίση πρέπει να τύχει συζήτηση και ήταν πολύ θετικό το ότι διοργανώσετε μια ε, εκδήλωση όπου ήταν παρόντες όλοι οι εμπλεκόμενοι. Δεν είναι ότι πηγαίνουμε εμείς στα κράτη-μέλη και του ζητάμε θέλουμε αυτό, εκείνο και εκείνο. Οι οργανώσει των κρατών μελών, σε τοπικό, σε περιφερειακό, σε οποιοδήποτε επίπεδο, πρέπει και αυτέ να υπομισθούν την ευθύνη του να αναπτύξουν τα δικά του επιχειρηματικά σχέδια για τέτοιου είδου θέματα και να προσπαθήσουμε να βρούμε μια προσέγγιση απόψεων για όλα αυτά τα θέματα μεταξύ μας. Αν υπάρχει λοιπόν ένα επιχειρηματικό σχέδιο από τις οργανώσεις αυτές, εμείς σίγουρα θα το αντιμετωπίσουμε με ευνοϊκό τρόπο και θα το λάβουμε υπόψη μας σε ό,τι αφορά τη δημιουργία ευρυζωνικών επικοινωνιών. Όταν μιλάμε για τις ε, επενδύσεις λοιπόν στην ευρυζωνική επικοινωνία και την διάδοσή της, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα σχέδια τα οποία προωθούν περισσότερη επένδυση στα θέματα αυτά. Μπορούμε επίσης να ενθαρρύνουμε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρηματοδοτήσει τέτοιου είδους ενέργειες. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία στο οπλοστάσιό μας. Δεν πρέπει λοιπόν να σταματήσουμε τις προσπάθειες μας προς την κατεύθυνση αυτή. και εγώ έχω τονίσει και ενώπιον σας και ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι και τα μικρά σχέδια και οι μικρότερες ευκαιρίες οι οποίες παρουσιάζονται μπορεί να είναι ιδιαίτερα πρόσφορες ακόμα και σε επίπεδο χωριών μπορούν να αναπτυχθούν υποδομές ευζωνικές και προσπάθειες για οικουμενική πρόσβαση στο ίντερνετ σε, στο χωριό αυτό που αναφέρω, στο οποίο αναφέρθηκα, στο Redland, οι κάτοικοι ανέπτυξαν το δικό τους δίκτυο με μια ε, επιχείρηση μέσα στο ίδιο το χωριό και το πιο ωραίο από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι είναι τρεις φορές ταχύτερο το ίντερνετ στο χωριό αυτό από ό,τι στο κέντρο του Λονδίνου. Αυτό για μένα είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, δεν πρέπει να περιμένει κανείς για πάντα. Θα μπορεί μερικέ φορές να βρει το δικό του δρόμο ο καθένας και τα κατάλληλα εργαλεία χρηματοδότησης για να αναπτύξει αυτήν την ε, ε, υποδομή. Θα επανέλθω τώρα και στο θέμα του, της χρήσης του ερτζιανού φάσματος. Η πρόταση της Κομισιόν έχει σαν στόχο σε ό,τι αφορά τις αδειοσυχνότητες να έχει το πρώτο πλαίσιο για στρατηγική σχεδίαση και εναρμόνιση της χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων και επομένω αναβάθμιση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τη υποστήριξη άλλων σημαντικών τομέων πολιτικής Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω είναι η προστασία του περιβάλλοντο, η υγεία, η δημόσια κτλ. Το ραδιοφάσμα είναι ένα σπάνιο δημόσιο πόρο. Θα το γνωρίζουμε αυτό και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συμβιβάσουμε τι ανάγκε όλων των τωρινών και ε, δυνητικών χρηστών με έναν τρόπο ο οποίο δεν θα οδηγεί σε διακρίσεις. Και να λάβουμε υπόψη όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική και πολιτιστική διάσταση της χρήσης του, του φάσματος ραδιοσυχνότητος. Χρειάζεται λοιπόν μια δημιουργική αντιμετώπιση και όχι να παραμείνουμε στο επίπεδο αυτού που είναι η παραδοσιακή χρήση του φάσματος, να μπορούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών με έναν τρόπο ο οποίος δεν οδηγεί σε διακρίσεις. Επίσης είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι δεν πρέπει να δημιουργήσουμε μια τεχνητή διάκριση μεταξύ της χρήσεως του ραδιοφάσματος για εκπομπές μονάχα, ενώ όλα τα υπόλοιπα πρέπει να καλύπτονται από ευρυζωνικές επικοινωνίες. Νομίζω ότι οι δύο αυτές μορφές επικοινωνίας ηλεκτρονικής μπορούν να έχουν μορφές συνέργειας και με το να τις συνδυάσουμε μπορούμε να αναπτύξουμε με φιλόδοξο τρόπο την ε, <clears throat> ψηφιακή διάσταση και να δώσουμε και περισσότερη δυνατότητα στην ευρωζωνική επικοινωνία, η οποία είναι εξέχουσας πολιτιστικής και κοινωνικής ε, σημασίας. Και οι περιοχές που δεν έχουν τέτοια πρόσβαση στα ευρωζωνικά προϊόντα έχουν ανάγκη να διατηρήσουν την πρόσβαση μέσα από το φάσμα ραδιοσυχνότητων. Δεν πρέπει να δούμε τα θέματα αυτά λοιπόν με ένα τρόπο ο, ο οποίος είναι απλοϊκός θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να χρησιμοποιηθούν από κοινού οι δύο αυτές δυνατότητες. Και εγώ έχω συζητήσει και με την Πρόεδρό σας και συμφωνώ απόλυτα με την άποψή σας ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες όλων αυτών των προσαρμογών. Γι' αυτό η Κομισιόν έχει δημιουργήσει τεχνικές επιτροπές οι οποίες επεξεργάζονται τα θέματα αυτά. Δεν έχω ακόμα τα πορίσματα τα τελικά αυτών των τεχνικών επιτροπών. Έχουμε και εμείς τους σοφούς μας στον τομέα αυτό, τους σοφούς τεχνικούς μας αν θέλετε και φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να προκύψει μια συμφωνία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω ζητήσει από όλους τους φορείς, όλους τους εμπλεκομένους να προωθήσουν καλύτερα πρότυπα στο μέλλον <clears throat> και επίσης να δημιουργήσουν και τεχνικές που ε, εμποδίζουν τις διακρίσεις ή τις θευλώσεις. Αν λοιπόν αυτό επιβεβαιωθεί εναπόκειται σε εμά να εφαρμόσουμε αυτά τα νέα πρότυπα και τις νέες τεχνικές στην νέα μαζική αγορά που δημιουργείται για τα προϊόντα ασύρματης ευζωνικής επικοινωνίας και η Κομισιόν παρακολουθεί τις διάφορες υπηρεσίες όπως είναι τα ασύρματα μικρόφωνα κτλ. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι κάποια από αυτά τα θέματα είναι εκτό τη δική μα αρμοδιότητα. Και η πρότασή μα υπογραμμίζει ιδιαίτερα την πολιτιστική και οικονομική σημασία αυτών των υπηρεσιών. Και βεβαίω ο στόχο μα είναι όχι μόνο να προστατεύσουμε αυτέ τι υπηρεσίε, αλλά να φροντίσουμε να έχουν και μελλοντική ανάπτυξη. Και αυτό είναι σημαντικό για να έχουμε πλούσιο περιεχόμενο στα μηνύε και βεβαίως να γεμίσουν οι μελλοντικοί διάδρομοι δεδομένων με περιεχόμενο το οποίο θα προσφέρει και λογικέ τιμέ. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα ζητήματα της, ε, του αισθήματο φάσματος γιατί διαφέρουν οι καταστάσεις από χώρα χώρα. Αλλά, όπως σας είπα, θεωρώ πως έχω δεσμευτεί ενώπιόν σας για το θέμα αυτό όμως. Ένα εργαστήριο που είχαμε στις 29 Οκτωβρίου πριν από 15 ημέρες μας βοήθησε να βρούμε κάποιες ε, μακροπρόσμες δυνατότητες για να βελτιωθεί η ενιαία αγορά για αυτό τον εξοπλισμό και τις υπηρεσίες. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας προς αυτή την κατεύθυνση. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να πω πως αναγνωρίζοντας πως ακόμα και αν το φάσμα είναι μια προτεραιότητα, είναι ένα ευρύτατο πρόγραμμα και βεβαίως ε, είναι ε, ένα ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει και θα έχουμε δαπάνες σε βάθος πενταετίας ε, και αυτό θα γίνει σε στενή συνεργασία με όλους και με εσάς και ξεκίνησα από εσά όχι γιατί είμαι ευγενική αλλά γιατί γνωρίζω την εξουσία που έχετε. Βεβαίω και τα κρατημέλη και ο κλάδος είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι χρήστε. Οπότε βλέπετε πως υπάρχουν πάρα πολλοί ενδιαφερόμενοι που πρέπει να διαβουλευτούμε μαζί τους. Οπότε αναμένω τη στήριξή σας για αυτό φιλόδοξο και σημαντικό πρόγραμμα. Θα ήθελα τώρα να αναφερθώ στο πρόγραμμα του 2011. Οι βασικές δράσεις για το επόμενο έτος και εδώ πέρα βέβαια προσπάθησα να επικεντρωθώ στα βασικά ζητήματα. Η ουδετερότητα του δικτύου, κάτι το οποίο είναι πολύ βασικό. Δημόσια διαβούλευση τελείωσε 30 Σεπτεμβρίου και όλες οι απαντήσεις έχουν δημοσιευτεί στο διαδίκτυο μας με την πρώτη αξιολόγηση από την Κομισιόν. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια σύνοδο κορυφής εδώ πέρα για να ακούσουμε όλους τους ενδιαφερόμενους και να προχωρήσει η συζήτηση η οποία ήταν πολύ χρήσιμη για μένα και ήμουν πολύ ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα της συζήτησης. Τώρα θα κάνουμε ένα απολογισμό και θα δώσω αναφορά σε εσάς και στο Συμβούλιο του Στομότερ Δυνατών για την ρύθμιση των τηλεπικοινωνιών πρέπει να αξιολογήσουμε πλήρως και δεν το λέω για πρώτη φορά τον αντίκτυπο και τις συνέπειες του κανονισμού περιαγωγής και θα σας πούμε τι θα προκύψει. Επίσης πρέπει να συζητήσουμε τι θα γίνει με τις διατάξεις για την καθολική παροχή υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ε, υπό το πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Αυτό είναι ένα από τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν. Αναμένουμε επίσης στο τέλος του επόμενου έτους μια νομοθετική πρόταση για να ενημερώσουμε και εσάς και το Συμβούλιο για την ε, επαναξιοποίηση της των πληροφοριών ε, του δημοσίου τομέα και υπάρχουν σημαντικές συνέπειες, ελπίζω όχι επιπλοκές, στον τομέα αυτών. Και επίσης θα ασχοληθούμε με ζητήματα που αφορούν την προσβασιμότητα του διαδικτύου. Κάθε Ευρωπαίος να είναι ψηφιακό σημαίνει για μένα ο κάθε Ευρωπαίος πραγματικά, άνθρωποι με αναπηρίες, οτιδήποτε. Κυριολεκτό δηλαδή ο κάθε Ευρωπαίος, κάτι το οποίο έχει σημαντικές συνέπειες για την κοινωνική συνοχή και για να διασφαλίσουμε πως η επανάσταση του διαδικτύου θα του συμπεριλάβει όλους. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τις προδιαγραφές προσβασιμότητας που πρέπει να είναι υποχρεωτικές για τα δημόσια site και να δούμε και τι θα γίνει με το σχέδιο δράσης για την αναπηρία που υιοθέτησε πρόσφατα η Κομισιόν. Επίσης θα δούμε τι θα γίνει με την εφαρμογή της οδηγίας για τις οπτικοακουστικές υπηρεσίες και οπωσδήποτε έχουν ευκαιρία να τα εξετάσω όλα αυτά μαζί σας του χρόνου με λεπτομέρειες, αλλά αυτά είναι κάποια από τα βασικά σημεία στα οποία θέλω να επιστήσω την προσοχή σας και βεβαίως θέλω να ακούσω τις αντιδράσεις σας. Το πρωί είχαμε το Συμβούλιο Πολιτισμού και εκπαίδευσης υιοθετήθηκαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Κληρονομιά και βεβαίω ελπίζουμε έτσι να δώσουμε περισσότερο βάρο στην ενημέρωση για τη σημασία της ευρωπαϊκής κινηματογραφικής κληρονομιάς κάτι το οποίο σημαίνει πως θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη νομική βεβαιότητα για να επιτρέψουμε σε αυτά τα θεσμικά όργανα να εκπληρώσουν την αποστολή τους προς το δημόσιο συμφέρον για την διατήρηση και την αποκατάσταση και την πρόσβαση σε αυτά τα έργα. Επίσης, προσκάλεσαν τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν πως ε, οι ταινιοθήκες ε, θα πρέπει να έχουν την δυνατότητα να υποφεληθούν από την μη εμπορική χρήση των ταινιών που υποστηρίζονται από εθνικά και περιφερειακά ταμεία και βεβαίως είχαμε και ανταλλαγές απόψεων ε, για τις ε, οπτικοακουστικές στοιχείες της ψηφιακή ατζέντα, ειδικά όσον αφορά τις προτεραιότητες των κρατών μελών και δυνατότητα να βελτιωθεί οριζόντια συνεργασία και συντονισμό σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Και βέβαια είχαμε και ένα γεύμα εργασίας ε, και με την Επιτροπή των Σοφών και έτσι να σας πω μεταξύ μας πως χαίρομαι για το ότι τρεις ενεργοί άνθρωποι αφιερώνουν τόσο χρόνο και προσπάθεια στο θέμα αυτό το οποίο του ζητήσαμε γνωρίζουμε πως το 3 είναι ένας συμβολικός αριθμός εν πάση περιπτώσει δεν πρόκειται για μια ομάδα ενδιαφερομένων πρόκειται απλά για άτομα, ελπίζουμε, με μια φρέσκια δημιουργική ματιά και είναι ενθουσιώδης μέχρι στιγμής δραστήριοι είχαν ταλέπονται όλες τις ευκαιρίες για κροάσεις, όπως ξέρετε επικοινωνία μαζί σας και τα λοιπά οπότε ό,τι ξέρετε ξέρω δεν έχουν ολοκληρώσει βέβαια το έργο τους. Και ό,τι μπορούν να κάνουν για να προετοιμάσουν την τελική έκθεση. Η οποία θα είναι, ελπίζουμε, συνεισφορά κλειδί για να αποφασίσουμε τις μελλοντικέ μας δράσεις σε σχέση με την ψηφιοποίηση και την Ευρωπαϊκή και νομίζω πως θα έχουν δυνατόν να ολοκληρώσουν το έργο τους και να μην κάνουν έτσι κομμάτια από εδώ και από εκεί. Αυτά έγιναν στη διάρκεια του γεύματος εργασίας με τους υπουργούς. Και εγώ πραγματικά έλαβα υπόψη πως στα βασικά συμφωνούμε όλοι. όλοι. Βεβαίω αυτό δεν προξενεί έκπληξη, ξέρετε ποια είναι τα βασικά, είναι και πολύ σημαντικά. Βεβαίω, μια που μιλάμε για το Συμβούλιο. Σε αυτή την περίπτωση ελπίζω να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ Νέλη. Αναφέρθηκε σε πάρα πολλά θέματα Λοιπόν, έχουμε κάποιους συναδέλφους που ζήτησαν τον λόγο. Κυρία Καμάεβα, η οποία είναι η συγγήτρια για την γνωμοδότηση για την πολιτική του φάσματος. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις πληροφορίες ε, που μας ε, δώσατε ως εισηγήτρια. Θα επικεντρωθώ στο πρόγραμμα για το ραδιοτηλεοπτικό φάσμα Νομίζω πως συμφωνούμε πως η ευρυζωνικότητα δεν έχει μόνο οικονομικό ενδιαφέρον αλλά και ενδιαφέρον από τη σκοπιά κοινωνικής και πολιτισμικής συμμετοχής. Δεν νομίζω να διαφωνούμε εδώ πέρα και δεν νομίζω να χρειάζεται να κάνουμε αυτή την τεχνητή διάκριση μεταξύ ίντερνετ και κλασικής τηλεόρασης. Και κλασικής τηλεόρασης. Εάν δούμε όμως τι προτείνει η Κομισιόν εδώ πέρα για το φάσμα, δεν είμαι τόσο αισιόδοξη, αντιθέτω ανησυχώ. Ειδικά στον τομέα της τηλεόρασης, αυτός είναι ο τομέας που μάλλον παραμελείται, γιατί λέει η ανακοίνωση της Κομισιόν πως σκέφτεται να πάει πέρα από τη δέσμη συχνοτήτων ε, των 800 κάτι το οποίο με ανησυχεί για το ότι το ζήτημα εδώ πέρα είναι η κλασική ραδιοτηλεόραση να φύγει τελείως από την επίγεια μετάδοση και ξέρετε πως έχουμε πολλούς αθμούς ιδιωτικούς ε, και δημόσιους που αποτελούν σημαντικό μέρος του πλουραλισμού και του πλουραλισμού των ΜΜΕ και χρειάζονται αυτές τις συχνότητες. Στη Γερμανία έχουμε τα χρήματα τα οποία επενδύθηκαν από τους ηλιοπτικούς σταθμούς στο ψηφιακό σήμα τα οποία θα πάνε χαμένα ξέρω. επίσης στη Γαλλία η επίγεια μετάδοση παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο από ότι σε άλλε χώρε δεν βλέπουν τόσο πολύ καλωδιακή και δορυφορική τηλεόραση και αν πάρουμε σοβαρά αυτό το οποία αποφασίσαμε στο πακέτο των τηλεπικοινωνιών, δηλαδή να έχουμε και πλουραλισμό και ποικιλία και βεβαίω να υπάρχει και ουδετερότητα ως προς τι τεχνολογίες τότε πρέπει να δούμε το ερώτημα μήπως, δεν ξέρω, δεν θα μιλήσω για ένα χώρο προστασίας, απλά να υπάρχει η δυνατότητα της επίγειας μετάδοσης για τηλεόραση και να μην κοιτάμε μόνο την οικονομική βιωσιμότητα. Θα πρέπει να γίνουν κάποιες επίσης βασικές διευκρινήσεις για το εάν θα μπορεί να συνεχίσει να μεταδίδεται με επίγειο τρόπο η ε, ραδιοτηλεόραση στην Ευρώπη. Επίση είπατε πως θα πρέπει να έχουν κάποιε αρμοδιότητε στα κράτη-μέλη. Συμφωνώ και εγώ εδώ πέρα γιατί ακριβώς οι διαφορές που υπάρχουν στα κράτη-μέλη οδηγεί, οδηγούν σε ότι χρειάζεται κάποια αυτονομία σε ένα συντονισμένο πάντα πλαίσιο. Αλλά και εδώ έχω την εντύπωση πως το πρόγραμμα του ραδιοτηλεοπτικού φάσματος δίνει περισσότερες αρμοδιότητες στην ε, Κομισιόν, τις οποίες παίρνει από τα κράτη-μέλη. Τελευταίο είναι βεβαίως το ζήτημα της επικάλυψης των συχνοτήτων, στο οποίο πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση, να μην οδηγηθούμε σε παρεμβολές και να δούμε βεβαίως... Ε, ε τι γίνεται και με τα σύρματα μικρόφωνα που είναι πάρα πολύ σημαντικά για οποιοδήποτε μικρό θέατρο να οδηγηθούμε σε ένα καθεστώς νομικής ασφάλειας ή τουλάχιστον να υπάρξει μία αποζημίωση για τις επενδύσεις οι οποίες έχουν γίνει γιατί ακριβώς στον τομέα αυτών της ε, πολιτιστικής επικοινωμορφίας θα πρέπει να δώσουμε το βάρος. Εντάξει, είναι καλή η οικονομική βιωσιμότητα αλλά δεν πρέπει να παραμελήσουμε και την άλλη πτυχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω ήδη στην, πει στην κυρία Κρούς ιδιωτικά ότι είμαστε ενωμένοι στον αγώνα για την πολιτιστική πολυμορφία. Το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι οποίοι παράγουν αυτά τα μικρόφωνα είχαν ήδη την έγκριση της Κομισιόν για να παραγάγουν αυτά τα μικρόφωνα και τώρα πρέπει να κάνουν κάποια αλλαγή. Γνωρίζουν όμως όλοι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και περιμένουν την ε, διαβούλευσή μας και τα, τα πορίσματά της. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Επίτροπε που ήρθατε να μιλήσετε στην Επιτροπή μας ε, και δέχεστε ερωτήσεις για να ακούσετε και τις απόψεις των μελών και να τις μεταφέρετε στην Κομισιόν, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το θέμα της ψηφιακή ατζέντα να μην το δείτε μόνο από την οικονομική και την τεχνική πτυχή, αλλά από την πολιτιστική που είναι σημαντικότερη. Η Πέτρα. Νομίζω, καλά είπε η Πρόεδρος πως μίλησε από καρδίες και είναι πράγματι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπε για το θέμα του φάσματος. Ε, κάτι το οποίο είναι σημαντικό τώρα για μένα. Η επέκταση του φάσματος ε, θα πρέπει βεβαίως να πάει προς την κατεύθυνση και της μετάδοσης δεδομένων, αλλά να δούμε και στην Ήπεθρο πώς θα οδηγηθούμε σε περισσότερη ευρυζωνικότητα ή, ή ευρυζωνικότητα. Μόνο μέσω του κινητού φάσματος ε, δεν ξέρω αν ε, επαρκεί μεσομακροπρόθεσμα γιατί οι τεχνολογικές δυνατότητες σήμερα δεν μας επιτρέπουν να μεταφέρουμε και μεγάλες ποσότητες ε, δεδομένων μέσω των συστημάτων κινητής. Οπότε θα έχουμε πάλι μειονεκτική θέση της υπαίθρου που είχαν μόνο παροχή μέσω των ασυρμάτων δικτύων. Δεν ξέρω τι έχει σκεφτεί η Κομισιόν για την Ήπεθρο. Θα μπορούσαμε να απλοποιήσουμε την παροχή οπτικών ε, ινών, αλλά έχω κάποια συγκεκριμένα ερωτήματα. Πώς ε, έχει η συζήτηση για τη νέα διαρθρωτική πολιτική μετά το 2013 και το δημοσιονομικό πλαίσιο, πόσα λεφτά έχουμε ή αν έχουμε. Γιατί ξέρετε το κόστος για την ε, επέκταση και της κινητής ευρυζωνικότητας αφενός είναι υψηλό, αλλά υπάρχει και η αναγκαιότητα παροχής ευρυζωνικότητας στους κατόχους της υπαίθρου για να μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν σε αυτά τα οποία προσφέρει το ίντερνετ ε, και από πλευρά πολιτιστική και από πλευρά επαγγελματική, οτιδήποτε. Πώς εκτιμάτε το κόστος ε, θα συμπεριληφθεί στο μέλλον της διαρθρωτικής πολιτικής και πώς βλέπετε τη στενή συνεργασία με το εθνικό και περιφερειακό επίπεδο έχετε κάποιες συγκεκριμένες ιδέες, κάποια ιδέα για το πώς θα μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε οικονομικά, γιατί ο πολιτισμός είναι πολύ σημαντικός, αλλά πρέπει να δούμε βέβαια και τι γίνεται με τη χρηματοδότηση και για το περιεχόμενο. Και άρα προκύπτει και ένα δεύτερο ερώτημα. Το θέμα της ουδετερότητας του διαδικτύου, το είπατε. Θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια πράγματα παραπάνω. Τι σκοπεύει να κάνει για να εγγυηθεί πως και στο μέλλον δεν θα υπάρχουν διακρίσεις στην πρόσβαση στο διαδίκτυο στο ευρωπαϊκό επίπεδο και είναι ιδιαίτερα σημαντικό κατά την άποψη της Επιτροπή μας το ίντερνετ να παραμένει στη διάθεση όλων εξίσου και ειδικά νομίζω αυτοί οι οποίοι είναι μικροί και προσφέρουν περιεχόμενο, αυτοί εξασφαλίζουν την ποικιλομορφία, την πολιτισμική. Δεν πρέπει να μείνουν σε μειονεκτική θέση πίσω από τους μεγάλους παρόχους που θα έχουν καλύτερες ταχύτητες στο ίντερνετ. Και άρα ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα εναντί των μικρών. Για μένα λοιπόν είναι σημαντικό να έχουμε πρόσβαση χωρίς καμία διάκριση και να δούμε πώς θα αναπτύξουμε εναλλακτικέ. χωρίς βέβαια να παίρνουν κάποιοι το ίδιο περιεχόμενο και να το ξαναπουλάνε, γιατί θα διηγηθούμε σε ολιγοπολιακές καταστάσεις, κάτι το οποίο ήδη έχει αρχίσει να συμβαίνει. «Ω Θεέ μου», λέει η πρόεδρος, «ελπίζω να τα να πρόλαβαν οι διερμηνείς». Θα δώσω και σε, άλλον, σε άλλη μια Γερμανίδα το λόγο, στην κυρία Τρίπελ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ, ον Γερμανίδα, θα μιλήσω στα αγγλικά. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Επίτροπο για την ομιλία της, κυρία Κρού, σας ευχαριστώ. Θέλω να υπογραμμίσω όλα αυτά που είπαν οι τρεις προηγούμενες ομιλήτρες από την Επιτροπή μας και να σας θυμίσω, να μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι στην πρώτη σας ομιλία για τις τηλεπικοινωνίες εδώ στην Επιτροπή μας μας είπατε ότι κατανοούσατε το ότι θα πρέπει να βρεθεί μια σωστή ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική πλευρά και στα πολιτιστικά θέματα. Τώρα που σας άκουσα για το θέμα των ραδιοφωνικών συχνοτήτων Βλέπω ότι ίσως να έχετε ξεχάσει το τι έχει κάνει μέχρι τώρα το Κοινοβούλιο στο πακέτο για τα Telecom. Εμείς μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει να περάσουμε ορισμένες τροπολογίες σε αυτό το πακέτο για τις τηλεπικοινωνίες και θα ήθελα παρακαλώ να λάβετε υπόψη σας σοβαρά αυτά τα οποία κάνει το Κοινοβούλιο. Δεν είναι σωστό να ξεκινάμε κάθε κοινοβουλευτική περίοδο εξ αρχής. Αυτά που κάναμε τα κάναμε με επικοδομητικό πνεύμα και ε, ίσως ε, ε, εφόσον τα ενσωματώσετε στην προσπάθειά σας να είναι ωφέλιμο για όλους. Μας είχατε υποσχεθεί ότι θέλετε εσείς να προσπαθήσετε να ισορροπήσετε την εμπορική οικονομική πλευρά με την πολιτιστική πλευρά. Αυτό πρέπει να σας το υπενθυμίσω. Όλοι ενδιαφερόμεθα φυσικά για την οικονομική επιτυχία των πραγμάτων, αλλά αυτά τα οποία συζητάμε, οι εκπομπές τις οποίες αναφερόμεθα, έχουν σχέση με την εθνοτική, την πολιτιστική ποικιλότητα και δεν είναι αυστηρά ένα θέμα οικονομικού ανταγωνισμού. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω λοιπόν αυτά τα οποία υπόθηκαν από την προηγούμενη ομιλήτρια. Από την άλλη μπορείτε να μας δώσετε κυρία Επίτροπε κάποιες, ερω... κάποιες απαντήσεις σχετικά με το διαδίκτυο. Δεν είναι μυστικό ότι στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ιδιαίτερα ανάμεσα σε εσάς και σε ε, άλλους επιτρόπους, υπάρχουν ορισμένες διαφορές σε σχέση με την ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς από τη μία και τις οικονομικές πλευρές που θα εμπεριέχει και από την άλλη θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή νέες μορφές απόδοσης κινήτρων σε δημιουργούς. Εφόσον μπορείτε σε αυτή τη φάση να μας πείτε τι συζητάτε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτό θα ήταν θετικό για μας. Ευχαριστώ κύριος Μπαρίς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Επίτροπος σίγουρα μας καθοδηγεί σε σωστές κατευθύνσεις σε σχέση με την προσβασιμότητα στο δίκτυο. Ε, στο... Θυμίζω ότι στο άμεσο μέλλον θα συζητήσουμε τέτοια θέματα και θα συζητήσουμε επίσης και τα θέματα της συνοχής. Χάρη στα διαρθρωτικά ταμεία, όταν ήμουν περιφερειακός υπεύθυνος στην Πολωνία, ήμουνα σε θέση να χρησιμοποιήσω τα ταμεία αυτά και να θέσω σε λειτουργία δίκτυα φάσματος. Αλλά είχαμε φυσικά το πρόβλημα των τελευταίων εκατοντάδων μέτρων όπου είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το τελευταίο κομμάτι να το καλύψει κανείς. Και σύμφωνα με αυτά τα οποία ζήτησε και η κυρία Τρούπελ θα ήθελα και εγώ να μου πείτε ποιος θα πρέπει να ηγηθεί αυτού του μοντέλου και ποιο είναι τελικά αυτό το μοντέλο το οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την πνευματική ιδιοκτησία όταν έχουμε να κάνουμε για πρόσβαση ε, σε ευρύτατη μορφή στο διαδίκτυο, σε έργα τέχνης, μουσική κτλ. Και τι είδους τεχνικές θα χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για να διασώσουμε θα έλεγα την πνευματική ιδιοκτησία για την ψηφιοποίηση τώρα του κινηματογράφου, των κινηματογραφικών έργων. Δεν είδαμε τίποτα στην ατζέντα την οποία προτείνεται. Νομίζω ότι η Ευρώπη εδώ έχει μείνει πολύ πίσω από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Θα πρέπει να είναι εφικτό για τους πολίτες ή οδήποτε βρίσκονται ε, να έχουν την δυνατότητα σε ψηφιοποιημένα κινηματογραφικά προϊόντα με την βέλτιστη δυνατή ε, ε, τεχνολογία μετάδοσης, όχι αναλογική φυσικά, αλλά ψηφιακή υψηλής ταχύτητας. Σχετικά λοιπόν με την ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών έργων και σχετικά με τα θέματα της μετάφρασης των υποτίτλων, είναι κάτι το οποίο είναι τμήμα μιας συγκεκριμένης γραμμής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα γίνεται άλλωστε μέσα από το πρόγραμμα Media λέει η Πρόεδρος. Δεν είναι αρμοδιότητα της κυρίας Κρούς. Αλλά καλό είναι να υπάρχουν θέματα τα οποία να συγκεντρώνουν την προσοχή δύο επιτρόπων ακόμα και αν τσακώνονται. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες. Η ευρυσονικότητα είναι το μέλλον και ε, του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και εσείς αποφασίζετε περισσότερα από τους υπουργούς πολιτισμού, αλλά μία πτυχή θα ήθελα να μάθω πώς την βλέπετε. Μιλάμε για την ανάπτυξη επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Έχουμε το πρόβλημα αυτό σε όλα τα έγγραφα και διαπιστώνω, παραδείγματο χάρη, στην κατάρτιση των δασκάλων, πως είναι ένα μεγάλο ένιγμα. Άρα επειδή μας, μας και η εκπαίδευση εδώ πέρα, αναρωτιέμαι γιατί δεν υπάρχει κατάρτιση των δασκάλων για τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Είναι παράδοση πως δεν χρειάζεται τίποτα. Βλέπει κανείς στα οπτικοακουστικά σε μία οθόνη. Αλλά σημαντικό είναι να μην ξέρουμε πως υπάρχει μόνο η τεχνολογία, αλλά και οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάτι με αυτή τη τεχνολογία, ίσως να το δουν κάπως κριτικά. Το λαμβάνετε αυτό υπόψη ή δεν έχει σημασία για εσάς και είναι εθνικό ζήτημα. Για τις επικοινωνιακές δεξιότητες. Όπως και οι προηγούμενοι συνάδελφοι θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα του περιεχομένου. Τι δυνατότητες επιλογών μπορεί να έχουμε σε σχέση με το περιεχόμενο. Πώς οι καλλιτέχνες οι οποίες θέλουν να συνεισφέρουν στην ψηφιακή τεχνολογία. Να αναφερθώ και στο θέμα της μετάβασης. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε τις μεθόδους μετάβασης από το ένα σύστημα στο άλλον. Ίσως το χρονικό διάστημα που έχουμε στη διάθεσή μας να είναι πάρα πολύ μικρό. και τι σχέσεις ε, μπορούμε να αποκαταστήσουμε με τις δημόσιες βιβλιοθήκες και τις βιβλιοθήκες μέσων ενημέρωσης γενικά που ελέγχονται από τοπικές αρχές. Ωραία, μπορούμε να κλείσουμε τώρα τη συζήτηση αυτή και έχει τη δυνατότητα η κυρία Επίτροπος να απαντήσει εφόσον το επιθυμεί. Η κυρία Τσουίπολ με έβαλε στη γωνιά. Εξετάτε βέβαια από το θέμα. Αν έχετε για μια στιγμή μονάχα την ιδέα ότι δεν παίρνουν στα σοβαρά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, πρέπει να σας πω αμέσως ότι δεν συμφωνώ. Αυτό δεν είναι λοιπόν σωστό. Υπήρξα και εγώ κοινοβουλευτικό στην προηγούμενη μου ζωή και είμαι συνηθισμένη στη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πια μετά από τόσα χρόνια. Επομένως, σας παίρνω απόλυτα σοβαρά. Αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε πάντα. Όχι. <clears throat> Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με την αντίληψη της σοβαρότητας κάνω ό,τι μπορώ πάντα για να αντιμετωπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τώρα θα ήθελα να δώσω μερικές απαντήσεις σε θέματα που είναι για μένα πολύ σημαντικά. Είμαι ευγνώμων λοιπόν για την ευκαιρία να τα συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Για τα θέματα του, των ραδιοσυγνωτήτων, του ραδιοφωνικού φάσματος. Αυτή είναι μια μοναδική πρόκληση που αντιμετωπίζει κανείς μια φορά στη ζωή του. Το γεγονός ότι είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε αυτή την ευκαιρία να αναδιαρθώσουμε τη χρήση του ραδιοφάσματος και γι' αυτό σας λέω ας επιταχύνουμε αυτές τις διαδικασίες. Υπάρχει ένα είδος κύκλου. Χρειάζεστε το ραδιοφάσμα για να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες ευρωζωνικής επικοινωνίας για να μπορέσουμε έτσι να εφαρμόσουμε την, το ψηφιακό θεματολόγιο. Και αυτό για πολλούς λόγους, είτε είναι οικονομική είτε είναι πολιτιστική είτε είναι εκπαιδευτική, όποιο και να είναι το επιζητούμενο. Πρέπει να κατανοήσουμε λοιπόν ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η δυνατότητα αυτή του ραδιοφάσματος για την ευζωνική επικοινωνία. Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε κατά πόσο αυτή η νέα ευκαιρία μας παρέχει αρκετό αρκετό τμήμα του φάσματος για να μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά τα οποία θέλουμε. Είναι προφανές ότι είμαστε φιλόδοξοι, ο καθένας έχει τη δική του προσέγγιση. Αλλά σε τελική ανάλυση θα πρέπει να καταλάβουμε πόσο φιλόδοξο είναι αυτό το πρόγραμμα. Όταν μιλάμε για το φάσμα για τις εκπομπές από τη μία πλευρά και την ευρυζωνική επικοινωνία από την άλλη πλευρά, δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα δεύτερο ψηφιακό μέρισμα η Κομισιόν είναι πεπισμένη, εγώ δεν πιστεύω στην αιώνια ζωή επί τη ευκαιρία, είναι η μία ευκαιρία σε μία ανθρώπινη ζωή και έχουμε μία σημαντική ευθύνη για το μέλλον και τις επερχόμενες γενναίες. Και έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι αυτή η ευκαιρία είναι πάρα πολύ σημαντική για να μπορέσουμε να διευθετήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Φυσικά παρακολουθούμε την κατάσταση. Θα ήταν ανόητο από τη δική μας πλευρά ότι <clears throat> ξέρουμε τι γίνεται και μπορούμε να κάνουμε τις απαραίτητες ενέργειες. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει η αποτελεσματική χρήση των ραδιοσυγνωτήτων. Βέβαια με την προϋπόθεση ότι εφόσον υπάρχει αρκετό ραδιοφάσμα το οποίο είναι διαθέσιμο πρέπει να χρησιμοποιηθεί προς το όφελος των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Και επειδή αναφερθήκατε στις ευκαιρίες που υπάρχουν για την ασύρματη ευρυζωνική επικοινωνία, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για κάτι τέτοιο. Εμείς αντιμετωπίζουμε τα θέματα των παρεμβολών με τους εμπειρογνώμονες και τους εμπλεκομένους, παρεμβολό στο ραδιοφάσμα δηλαδή, και συζητούμε κατά πόσον υπάρχουν δυνατότητες να έρθουν, αν θέλετε μπορούν να έρθουν και οι εμπειρογνώμονες μας για τα θέματα αυτά να έρθουν να σας εξηγήσουν ακριβώς περί πρόκειται. Νομίζω ότι ο επικεφαλής των, ο αρμόδιος γενικός διευθυντής μπορεί να τα παρουσιάσει αυτά πλήρως. Έχω πάντως την υποστήριξη των εμπειρογνωμόνων και των εμπλεκόμενων για τα θέματα αυτά. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είμαστε επάγρυπνοι. Για τα κράτη-μέλη τώρα. Θα πρέπει να προβλέψουν και ποιε είναι οι οικονομικές επιπτώσεις βάσει των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και διακινδυνεύω εδώ πέρα, θα έλεγα ότι το πρόβλημα αυτό με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πρέπει να επιληθεί. Και στο Συμβούλιο μιλώντας για το θέμα των κινηματογράφων, με πληροφορήσανε ότι τα μικρά, οι μικροί κινηματογράφοι οι οποίοι περνούν σε ψηφιακές προβολές υπάρχει χρηματοδότηση μέχρι 75.000 ευρώ. Νομίζω ότι αυτό θα ευνοήσει την επίτευξη λύσεων. Είναι πολλοί λοιπόν οι οποίοι γνωρίζουμε αυτά τα προβλήματα και πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν θύματα αυτής της μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο. Και στις περιοχέ υπαίθρου η χρήση της ασύρματης επικοινωνίας για τις ευρυζωνικέ υπηρεσίες είναι κατά την άποψή μα η καλύτερη λύση σε πάρα πολλέ περιπτώσεις. Άμα δείτε την έκταση του σταθερού δικτύου επικοινωνιών βλέπετε ότι δεν είναι βιώσιμη η χρήση του από οικονομική έποψη. Επομένως, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι υπάρχει μονάχα ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο μας, ένα εργαλείο μονάχα για την επικοινωνία. Υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την ευζωνική επικοινωνία και την ασύρματη και τους δορυφόρους. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι κάνουμε την βέλτιστη χρήση όλων αυτών των δυνατοτήτων, ώστε οι πολίτες αυτής της περιοχής δεν θα υπολείπονται σε δυνατότητες επικοινωνίας. και μας ενδιαφέρει όλοι, είτε είναι σε ύπεθρο, είτε είναι ε, σε απομονωμένες περιοχές, θα πρέπει να έχουν κάλυψη από, επικοινωνία, από επικοινωνιακή πλευρά. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε τις τεχνολογίες οι οποίες είναι διαθέσιμες και αυτές είναι και οι περιοχές όπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν επωφελώς οι κρατικές επιδοτήσεις και, τα, τα, και το Περιφερειακό Ταμείο για την επέκταση του δικτύου του ευρυζωνικού. η ουδετερότητα του δικτύου. Αυτό είναι ένα συναρπαστικό θέμα. Εγώ λέω πάντα όταν υπάρχει μια συζήτηση για την ουδετερότητα του ίντερνετ και των δικτύων μάλλον, ότι πρέπει να έχουμε μια σαφήνεια για το τι λέμε, τι εννοούμε όταν μιλάμε για ουδετερότητα. Αν συγκριθούμε με τις Ηνωμένε Πολιτείες, αυτό είναι δύσκολο να κάνουμε μια σύγκριση, είναι πολύ διαφορετικές οι Ηνωμένε Πολιτείες και είναι διαφορετικός ο ανταγωνισμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ας παραμείνουμε λοιπόν στα δικά μας ευρωπαϊκά αυγά, όπου και εκεί υπάρχει ανταγωνισμός. Με ενδιαφέρει να είναι ανοιχτή η πρόσβαση στο ίντερνετ και να υπάρχει δυνατότητα επιλογής των καταναλωτών. Αυτό διακυβεύεται. Αυτό τουλάχιστον εγώ θέλω να τονίσω και να προωθήσω. Να υπάρχει ανοιχτή πρόσβαση, ανταγωνιστική πρόσβαση, να υπάρχουν πολλαπλές λύσεις για τον καταναλωτή ώστε να υπάρχει η δυνατότητα επιλογής. Μετά χρειάζεται και μια συνεκτικότητα ή θα δώσουμε επιλογή στον καταναλωτή και τότε θα είναι ανοιχτή η πρόσβαση και όλα αυτά δεν είναι δωρεάν γεύμα. Δεν σημαίνει ότι η ελεύθερη πρόσβαση δεν σημαίνει ότι δεν θα τιμολογούνται οι υπηρεσίες οι οποίες δίνονται στον καταναλωτή. Πρέπει λοιπόν να τονίσω και ότι η απελευθέρωση του φάσματος δίνει περισσότερες ευκαιρίες στον καταναλωτή. Γι' αυτό θα έπρεπε να είμαι ανόητη για να μην καταλάβω ότι και για σας αλλά και για την Κομισιόν είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το φάσμα. Και σε τελική ανάλυση η Κομισιόν ουσιαστικά ενσωμάτωσε και απεδέχθη τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. εξάλλου, το πακέτο μας αναφέρεται, ε, αναφέρει όλα αυτά με μία γλώσσα η οποία είναι πιστεύω εύληπτη και κατανοητή. Οι εκπομπές ε, υπάρχουν πολλές δυνατότητε, υπάρχει και η χρήση του ίντερνετ και αυτό το αναγνωρίζουμε με την πολιτική μας περί ραδιοσυχνοτήτων. Ε, εάν έχετε αμφιβολίες παρακαλώ πέστε μου που διαφωνείτε. Η γλώσσα του σώματός σας δεν μου δίνει την εντύπωση ότι συμφωνείτε απόλυτα μαζί μου, αλλά θα έλεγα ότι αν έχετε αμφιβολίες, πέστε μου και αφήστε με να γνωρίζω ποια είναι η θέση σας. Πνευματική διοκτησία και το σενάριο το οποίο υποστηρίζουμε εμείς. <clears throat> Εμείς θέλουμε ένα σενάριο, υποστηρίζω ένα σενάριο, όπου οι καλλιτέχνες και οι χρήσεις, χρήστες θα λαμβάνονται υπόψη. Όταν μιλάμε για τους παραγωγούς και τους ε, πνευματικούς δημιουργούς αξίζουν αμοιβή για τις υπηρεσίες τους και πρόσθετες αν χρησιμοποιούνται σε ψηφιακό επίπεδο <clears throat> και θα πρέπει να έχουμε μια καλύτερη αίσθηση για τα θέματα αυτά. Παραγωγή, χάρη περίπτωση της μουσικής οι δραστηριότητες κατεβάσματος μέσα σε εισαγωγή από το ίντερνετ διακυβεύονται αυτή τη στιγμή. Και η ψηφιακή ενιαία αγορά μπορούμε να πούμε ότι λειτουργεί στην Ευρώπη. Δεν ήταν τόσο δύσκολο να επιτύχουμε ότι έχουμε φτάσει σε μια τέτοια αγορά. Τώρα, το κατέβασμα πνευματικών προϊόντων είναι παράνομο. Ως πολιτικός Νομίζω ότι εσείς πρέπει να αντιμετωπίσετε το θέμα αυτό. Αν θεωρείτε ότι κάτι είναι παράνομο θα πρέπει να δράσουμε. Ξεκινά τώρα η συζήτηση. Στρεφόμαστε εναντίον της πειρατείας, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό δεν σημαίνει αυτό ότι αυτό είναι επαρκές αφ' αυτού. Θα πρέπει να εστιάσουμε στην συστημική προσέγγιση. Και θα πρέπει να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας. Έχουμε ένα σενάριο το οποίο είναι, γίνεται από δύο πλευρές. Πρέπει να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι οι πνευματικοί δημιουργοί θα την χάνουν της απαραίτητης αμοιβή, ώστε να μπορούμε να περιμένουμε και περισσότερα πολιτιστικά προϊόντα από αυτούς. Αλλιώς τους χάνουμε. Θα πάνε σε μια άλλη δουλειά όπου θα πληρώνονται Καλύτερα μεν, αλλά εμεί δεν θα απολαμβάνουμε τα πνευματικά του προϊόντα. Γνωρίζει λοιπόν η Κομισιόν και ο Μισελ Μπαρνιέ το γνωρίζει και εγώ το ξέρω. Και ο Μισελ είναι ο πρώτο ο οποίο εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Πολλέ φορέ είναι αρνητικά τα πράγματα, άλλε φορέ είναι θετικά. Αλλά το ψηφιακό θεματολόγιο είναι ένα οριζόντιο κατάλογο πρακτέου για την Κομισιόν και για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν δεσμευτεί προς την κατεύθυνση αυτή. Επομένως, δεν είναι ότι άλλαξα άποψη, δεν μου αρέσει κάτι, δεν το θέλω κτλ. Όχι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξασφαλίσουμε το ταχύτερο δυνατό, γιατί ο χρόνος από μόνος του δεν θα λύσει όλα τα προβλήματα όσο πανδαμάτων και να είναι. Και γι' αυτό ανησυχώ και για το θέμα του κατεβάσματος από το ίντερνετ, και υπάρχουν πολλοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα αυτά, αυτό. Κάποιος ο οποίος ασχολείται για αυτό το θέμα μου είπε ότι χάνουμε μια ολόκληρη γενιά. Γιατί εμπλέκονται οι νέοι σε αυτή τη δραστηριότητα που δεν κάνει εύκολη τη δουλειά των καλλιτεχνικών δημιουργών. Η ηλεκτρονική μάθηση και η ηλεκτρονική ο ηλεκτρονικός αλφαβητισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό της ψηφιακής ατζέντα του ψηφιακού θεματολογίου. Σημαντικό για τους μαθητές, για τους νέους, για τους φοιτητές να έχουν την ικανότητα να πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι μαθητές και οι φοιτητές να αποκομίζουν την ψηφιακή πληροφορία. Αλλά αν δεν, το έχουν, δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και οι διδάσκοντες, αυτό δεν θα οδηγήσει πουθενά. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν και σε εθνικό επίπεδο τις ευθύνε που έχουν όλοι αυτοί σε επίπεδο εκπαιδευτικό και να πείσουμε όλους τους υπουργούς που εμπλέκονται σε διάφορες πτυχές της ε, ψηφιακής ατζέντα, να τους πείσουμε να δράσουν το ταχύτερο δυνατό και εξάλλου είναι συναρπαστικό, είναι εγωιτευτικό όλο αυτό. Επισκέφθηκα ένα σχολείο σε μια φτωχή περιοχή που είχαν εξοπλισμό ψηφιακό και ήταν πολύ καλά εκπαιδευμένοι και οι καθηγητές τους για τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων και έκανα τη δουλειά τους με ενθουσιασμό και πάθος και μου δείξανε μετά από την επίσκεψή μου το γεγονός ότι οι παππούδες και οι προπάποι των παιδιών ερχόντουσαν στο σχολείο να μάθουν ένα-δύο πράγματα γιατί τα παιδιά τους τους εδίδασκαν σύμφωνα με το σύνθημα «Γυράσκω αίδιδασκόμενος». Κάποιοι από αυτούς είχαν προχωρήσει τόσο πολύ που θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και, και επιχειρηματικές δραστηριότητες. Και είπαμε ναι θα το αντιμετωπίσουμε και εμείς αυτό. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο μου δίνει έναυσμα να συνεχίσω σε αυτό το τόσο συναρπαστικό θέμα και προσβλέπω στην εφαρμογή αυτών των ενεργειών. Uh, πρέπει λοιπόν να... Θα πρέπει να προσέξουν όλοι αυτά τα οποία είπαμε και οι κινήσεις ε, ε, αυτών που σας ε, άκουγαν δεν ήταν αρνητικές επειδή δεν πίστευαν αυτά που λέγατε αλλά επειδή πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί και να συνειδητοποιήσουμε ότι ορισμένα πράγματα δεν μπορούμε να ανταλλάξουμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Του χρόνου το αργότερο θα τα ξαναπούμε. Απευθύνομαι τώρα λοιπόν στην Μαντλέν, τη Γενική Διευθύντρια, να μας πει τι θα γίνει εδώ πέρα από τεχνική σκοπιά με αυτά τα οποία είπαμε για να μην παραμελήσουμε μετά του πολιτισμού. Ευχαριστούμε, Νέλη. Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ε. so I hope that you... Ελπίζω να τα βρείτε λοιπόν. Ευχαριστώ πολύ και γεια σας. Περνάμε στο σημείο 9, δεν έχει μείνει και κανείς. Ευρωπαϊκό έτος ενεργού γύρωσης. Ναι, ου, εδώ. γυρνάμε μαζί. Καλά τα λέτε. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. οπωσδήποτε είναι αλήθεια πως γυρνάμε Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται ε, στην ηλικία μου και στην εμφάνισή μου το ότι είμαι εισηγητής για αυτή την έκθεση. Του Σάββατο είναι και τα γενέθλιά μου, 47 ετών θα γίνω, κάποιοι θεωρούν πως είναι έτσι μια αξιοσέβαστη ηλικία αυτή για έναν άντρα. Ε, εν πάση περιπτώσει θα προσπαθήσω να το ξεπεράσω. Κυρία Πρόεδρε, η γύρανση αυτή ή ενεργός και η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι κάτι το σημαντικό και ειδικά για το 2012. Ο Μάρτιν Κάστλερ είναι επικεφαλής εδώ πέρα η συγητής Είναι ένας νεότατος όμως άντρας τώρα βγάζει τις πρώτες ε, άσπρες τρίχες, αλλά κάτι έχει αυτός να μας πει για τη γύρανση. Ανακαλύψαμε ότι δεν υπάρχει προπολογισμό γι' αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Δεν ότι χρειαζόμαστε και πολλά λεφτά, αλλά γεγονό είναι πως αν είναι να εργανώσουμε το ευρωπαϊκό έτος αλληλεγγύης των γενεών, καλό είναι να κάνουμε και καμία εκδήλωση για να το καταλάβει κανείς. Αλλιώς δεν καταλαβαίνει ο κόσμος ότι υπάρχουν αυτές τις θεματικές χρονιές. Είμαι σίγουρος λοιπόν πως ο κύριος Κάστλερ θα φροντίσει να εμφανιστεί μια γραμμή στον προπολογισμό. Και το υποστηρίζουμε. Καλό θα είναι να κάνουμε έτσι μια ωραία εκδήλωση, να συζητήσουμε αυτό το θέμα δημοσίως. Είναι και επίκαιρο Εάν δείτε τις προσεχείς συζητήσεις για την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης σε πολλές χώρες, όπου μιλάμε για την ε, σταδιακή συνταξιοδότηση της μεταπολεμικής γενιάς, ε, του baby boom, άνθρωποι που έχουν πολλές γνώσεις, οι οποίες αποσύρονται από τον κόσμο της εργασίας και καλό θα ήταν να τις έχουμε, ακόμα και όταν βγουν στη σύνταξη. Όλα αυτά, όλη αυτή η εμπειρία αυτών των ανθρώπων που δεν πρέπει να τη χάσει η κοινωνία πρέπει να φροντίσουμε στο μέλλον η... τα γυρατιά να είναι αξιοπρεπή. Στην καταναλωτική μας κοινωνία βεβαίως ε, έχουμε την εντύπωση πως μόνο η εσωτερική αγορά μετράει και όσοι συνεισφέρουν στην εσωτερική αγορά έχουν σημασία και οι υπόλοιποι να πάνε να πνιγούνε τα παιδιά πάμε στα ιδρύματα, τους γέρους πάμε στα ιδρύματα, τους ανάπηρους στα ιδρύματα. Οι μόνοι που αξίζουν να ζουν σε αυτή την κοινωνία είναι αυτοί που είναι από τα 20 έως τα 55. Δεν είναι σωστό αυτό. Όλοι έχουν την ατομική τους αξία, αξιοπρέπεια, τη ζωή τους. Οπότε η γύρανση είναι κάτι το πολύτιμο. Είναι δώρο το να μπορεί κανείς να μεγαλώνει και αν γίνει αυτό με έναν τρόπο που θα τους επιτρέπει να εκμεταλλευτούν το σώμα και το πνεύμα τους τόσο το καλύτερο. Βεβαίω θα δώσουμε και έμφαση στη διαβίου μάθηση και τον αθλητισμό. Ξέρουμε Έχουμε και το σχετικό σεμινάριο. Ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμό. Νου υγιή, τη υγιή. Πρέπει επίση να αναφέρουμε πω το ότι είναι κανεί ηλικιωμένο δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να μαθαίνει. Γυράσκο αή δασκόμενο. Επίσης υπάρχει το θέμα της εθελοντική εργασίας. Έχουμε πολύ ικανούς ανθρώπους ηλικιωμένους, ικανούς από όλες απόψεις και σωματικά. Δεν λέω να τους εκμεταλλευτούμε, αλλά μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα για την κοινωνία. Πρέπει να συνεισφέρουν και πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να τους... για να εμπλακούν. Ε, έτσι θα αναδιανεμηθεί η γνώση από τη μία γενιά στην άλλη. Δεν ξέρω τι γίνεται στις άλλες χώρες αλλά στη Φιλανδία, δηλαδή όταν ήμουν εγώ μικρό παιδί λέμε τώρα, τα Σαββατοκύριακα πηγαίναμε στα γήπεδα και υπήρχαν μεγαλύτεροι άνθρωποι με το χρονόμετρο και μετρούσαν τις επιδόσεις μας. Ihmiset, jotka lähtevät mukaan tuommoiseen urheiluseuratyöhönkin tai nuorisoseuratyöhön tai muuhun tämän tyyppiseen vapaaehtoistoimintaan. Τώρα, μα πάει κανείς στο γήπεδο και σωστοί όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα σκέφτονται μόνο πόσα θα βγάλουν, εάν θα πληρωθούν. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά χρήσιμα πράγματα που μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι εθελοντικά στην Ευρώπη. Το χρήμα δεν φέρνει την ευτυχία. Αν δώσει κανείς ο χρόνο του εθελοντικά μπορεί να κερδίσει. Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε πως επειδή εξελίσσεται τόσο γρήγορα η τεχνολογία καθώς ε, προκύπτουν ε, νέες τεχνολογίες πρέπει αυτό να γίνεται με τρόπο ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν και οι νέοι για οι ηλικιωμένοι. Όλα τα στρώματα της κοινωνίας ανεξαρτήτως φύλου ηλικίας πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν στην τεχνολογική πρόοδο και θεωρώ πως η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών έχει ένα ρόλο να παίξει εδώ πέρα. Κύριε Πρόεδρε, παρά το ότι θα ολοκληρώσουμε σε 6,5, εγώ θα ολοκληρώσω τώρα. Λοιπόν, χρειαζόμαστε λεφτά, χρειαζόμαστε μια γραμμή του προπολογισμού για την πρόθεση της ενεργού γύρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Χρειαζόμαστε εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, να προσελκύσουμε την προσεχή στα ζητήματα αυτά, πολιτιστικά, αθλητικά και να είναι διαθέσιμα όλα αυτά στους ηλικιωμένους να τονίσουμε τον ε, εθελοντισμό και θα το λέμε συνέχεια και θα πρέπει βεβαίω να είναι διαθέσιμο αυτό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Αυτά κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ και θέλω να ακούσω βεβαίω και τις ερωτήσεις ε, των συναδέλφων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ Χάνου. Όλοι. Έχουμε καταλάβει ότι πέρασε από τον κουρέα σου πρωτού έρθεις εδώ να μας κάνεις αυτή την παρουσίαση. Λοιπόν, η κυρία Σάλτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να πω καταρχάς ότι εξπροσωπώ τις απόψεις της σκιώδους εισηγήτριας κυρία Σερανόβα που δεν είναι δυνατόν να είναι ανάμεσά μας σήμερα. Και εγώ στην Ιρλανδία έχω ασχοληθεί πάντως με τα θέματα αυτά και θεωρώ ότι είναι μια προτεραιότητε για τα επόμενα δέκα χρόνια. Το ότι γερνάει η Ευρώπη είναι αντικείμενο πολλών συζητήσεων ο μέσος όρος των Ευρωπαίων πολιτών αυξάνεται και ταυτόχρονα οι αριθμοί γεννήσεων έχουν αρχίσει να μειώνονται. Να σας παρουσιάσω κάποια στοιχεία της ε, Eurostat. Από το 2012 ο ενεργός πληθυσμός θα αρχίσει να μειώνεται σημαντικά. Ο πληθυσμός άνω των 60 θα αυξηθεί ανά 2 εκατομμύρια ανά 2 έτη Σήμερα είναι 85 εκατομμύρια οι άνω των 60 και θα φτάσουν τα 150, ε, τα 150 εκατομμύρια το 2060. Το προσδόκιμο θα αυξηθεί ε, κατά 8 χρόνια και τα στοιχεία αυτά προέρχονται από έγγραφα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως επίσης και των Ηνωμένων Εθνών. Η χάρτα λέει ότι είναι καθήκον μας να βοηθήσουμε τους ηλικιωμένους να ζήσουν τη ζωή τους μέσα στην αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη και πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενιές. Η στρατηγική του 2020 υπογραμμίζει τη σημασία της αλληλεγγύης αυτής για την κοινωνική συνοχή στην κοινωνία. Οι ηλικιωμένοι δεν είναι απλά θα έλεγα κάποια στοιχεία τα οποία φεύγουν από την αγορά εργασίας αλλά παίζουν σημαντικό ρόλο στους κοινωνικούς κύκλους, τους οικογενειακούς, τους φιλικούς, τους επαγγελματικούς και τους καθιστά είτε με θελοντικό τρόπο είτε με την απλή φυσική τους παρουσία σημαντικά στοιχεία. ένα 60% βοηθούν τις οικογένειές τους ενεργά, 12% βοηθούν εκτός των οικογένειών σε διάφορες κοινωνικές αποστολές. Και αυτό ορίζεται ακριβώς σαν δραστήρια τρίτη ηλικία. Αυτό δεν δείχνει μόνο τις δυνατότητες αλλά και τα εμπόδια τα οποία αντιμετωπίζουν. Στην Ευρώπη όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω της ηλικίας τους για λόγους υγείας κυρίως. Έχουν προβλήματα επίσης στην πρόσβαση νέων τεχνολογιών. Η απασχολησιμότητα αυτών που είναι 55 με 64 αυξήθηκε τα τελευταία χρόνια από 37 σε 46%. Αυτός ήταν ένας από τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας. Από την άλλη, οι διακρίσεις και η πρόσβαση σε σημαντικές υπηρεσίες ε, γίνεται πιο σημαντική. Η γύρανση έχει επίσης και άλλες πλευρές. Το 22% των γυναικών και 16% των ανδρών ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Εδώ δεν έχουμε βρει τις κατάλληλες λύσεις. Για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς, όπως είπε και ο, ο μιλητής, είναι η χρηματοδότηση. Αυτό είναι θέμα αρμοδιότητα των κρατών μελών αλλά μέσω των μειώσεων των προϋπολογισμών και των εξοικονομήσεων δαπανών έχουν μειωθεί οι παροχές των υπηρεσιών εις βάρος των παλαιών γενεών. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να παίξει το ρόλο του συντονιστή ε, σε διάφορα επίπεδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να θέσει σε λειτουργία πολιτικές που να επηρεάζουν θετικά τη ζωή των ηλικιωμένων. Οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες πρέπει να εμπλακούν επίσης διότι εκεί παρέχονται οι υπηρεσίες του ηλικιωμένου και ακριβώς εκεί θα μπορέσει να παίξει ρόλο και το ευρωπαϊκό έτος. Ευχαριστώ να σας υπενθυμίσω ότι δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι επί της ουσίας. Εμείς αντιμετωπίζουμε μονάχα τις πολιτιστικές πλευρές και τις πλευρές εκπαίδευσης. Πρέπει λοιπόν στις προτάσεις μας να δείξουμε κάποια αυτοσυγκράτηση. Αλλά πραγματικά χάρη για θέματα ε, διαβίου ε, μάθησης είμαστε εμείς που είμαστε αρμόδιοι. Ο Πόρης έχει το λόγο λοιπόν. Ως επόμενος ομιλητής ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσο πιο γρήγορα κατανοήσουμε ότι γερνάμε, τόσο καλύτερα η δημογραφική αλλαγή έχει μία αδηρητότητα. Η παιδεία είναι σημαντική. Τώρα υπάρχει πανεπιστήμιο της τρίτης ηλικίας. Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι αυτά τα ιδρύματα, πόσο προσιλωμένοι στο ρόλο τους είναι τα πανεπιστήμια της τρίτης ηλικίας και μπορούμε σίγουρα να ανταλλάξουμε βέλτιστες πρακτικές στην Ευρώπη. Επιπλέον, η ενεργός χείρανσης παρά την συνταξιδότηση. Όλοι θέλουν να συνεχίσουν να εργάζονται και παρά την συνταξιδότησή τους. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο προς όφελος των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να συνεχίζουν να εργάζονται με μερική απασχόληση ή με απασχόληση τριών τετάρτων, χάνουμε ευκαιρίες. Έχουμε επίσης την εθελοντική εργασία που μπορούν να κάνουν αυτοί οι ηλικιωμένοι. Θα πρέπει να σπάσουμε όχι τι αλυσίδε, αλλά τα στερεότυπα. Η Βουδαπέστη είναι γνωστή για τα ε, ιαματικά της λουτρά και για τα μπαρ που έχει. Ξέρετε ότι αυτά ανέρχονται στην εποχή των Ρωμαίων. 90% των ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτά τα ε, η αματικά λουτρά μέχρι το απόγευμα είναι 80 με 90 ετών. Με τις καλές πρακτικές, αν έχετε κάτι το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, μπορούν να μεταλαμπαδευτούν αυτά τα παραδείγματα. Ο κύριος Σκέλη. Ευχαριστώ, ρε κύριο Σκέλη. Αμικρόφωνος όμως. Σύντομος θα είμαι. Γιατί νομίζω ότι οι άλλοι ομιλητές έχουν καλύψει τα περισσότερα θέματα που ήθελα να πω σε σχέση με τη γύρανση. Θέλω να τονίσω ότι για μένα είναι κρίμα <clears throat> ότι δεν έχουμε μια γραμμή του προπολογισμού που να αντιμετωπίζει αυτό το θέμα παρά τις συζητήσεις που είχαμε στο παρελθόν. Και εκφράζουμε μονάχα πόθους, ευσεβείς και όχι πρακτικές λύσεις. Ενώ υπάρχουν πολλοί τρόποι υποστήριξης της Ενεργού γύρανση, ιδίως το όλο θέμα της διαβίου για τους ηλικιωμένου. Πολλοί άνθρωποι, πάνω από τα 60 τους, έχουν τις απαραίτητες γνώσεις για τους υπολογιστές. Θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τις δυνατότητές τους, αν μπορούμε να έχουμε καλύτερα εργαλεία τα οποία τους επιτρέπουν, παραδείγματος χάρη, να κλείνουν πτήσει στο διαδίκτυο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να δούμε αυτό. Επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε καλύτερα μορφές μεταβατικής συνταξιοδότησης. Αλλά θα χρειαστούμε να έχουμε και χρηματοδότηση στο προπολογισμό, μια γραμμή του προπολογισμού για αυτό. αυτά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θα ήθελα να δώσω μια σειρά που παρατηρήσα από τη δική μου πλευρά. Εγώ έχω διατυπώσει ότι χρειαζόμαστε αυτό που λέμε senior service. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι φτάσαν στην ηλικία της συνταξιοδότησης θα πρέπει να είναι έτοιμοι να υπηρετήσουν την κοινότητα στην οποία ζουν. Ιδίως σε χώρες που χρειάζονται τη βοήθειά τους. Χώρες όπως είναι η Βοσνία Ζεγοβίνη, όπως είναι το Κοσφοπέδιο, να βοηθήσουν τους νέους να ανοικοδομήσουν τις χώρες τους. Υπάρχουν πολλές τέτοιες δυνατότητες χώρες στα ανατολικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουκρανία, Αζερβαϊτζάν, Μολδαβία. Υπάρχουν τόσες δυνατότητες. Υπάρχουν πάρα πολλοί μηχανικοί παγκοσχάροι χάρη οι οποίοι μπορούν να πάνε σε αυτά τα μέρη μετά στη συνταξιοδότησή τους αντί να κάθονται και να παίζουν το κομπολόι τους. Δυστυχώς αυτή η έννοια του senior service δεν έχει ακόμα εισέλθει στο πνεύμα της Κομισιόν. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε με τη βοήθεια της δικής μας Συμβολήσει στα θέματα αυτά να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να αναφέρω. Η Κομισιόν είναι παρούσα, αλλά θέλω να του πω ότι είμαστε ακόμα σε επίπεδο πρώτη συζήτηση. Όταν έχουμε ένα έγγραφο εργασία, θα είναι πολύ πιο εύκολο να πάρει θέση η Κομισιόν για τα θέματα αυτά. Είναι η πρώτη φορά αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σα. Ο αγαπητό Χάνου Τάκκουλα έχει το λόγο για να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ξέρω πως... Ήξερα πως θα έρθω να μιλήσω για τη γέναση, οπότε είπα να φτιαχτώ λίγο. Αλλά συνειδητοποιώ πως και η σκιώδη συγκήτρια πέρασε από το κομμωτήριο. Είναι κρίμα το ότι δεν εντυπωσιάσαμε περισσότερους. καμιά φορά... Καμιά φορά δίνουμε και τα 23 ε, ευρώ στο κομμωτήριο και πάνε χαμένα γιατί δεν μας βλέπει κανείς. Οπότε ευχαριστώ τους συναδέλφους οι οποίοι Φανίστελρη και Κασλή να προσθέσω στον τίτλο και αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. δεν ξέρω. Νομίζω ότι θα γίνονταν έτσι πολύ σχηνοτενής ο τίτλος. Καμιά φορά καλό είναι έτσι να είναι μικρός. Σωστά είπε η Πρόεδρο πω πρέπει να εστιαστούμε στον τομέα του πολιτισμού και εγώ προσπαθώ να περιοριστώ εκεί πέρα. Ο Κάστλερ κάλυψε τα ζητήματα τη απασχόληση, δημογραφική αλλαγή τα επόμενα 50-60 χρόνια. Οπότε προσπαθήσουμε να μείνουμε εντός της εντολής μας. Δηλαδή εκπαίδευση, πολιτισμός, αθλητισμός. Οι ιδέες μου δώσατε είναι μια πολύ καλή αρχή. είμαι σίγουρος πως με το να αρχίσω να γράφω θα γεράσω έτσι και με πιο αξιοπρεπή τρόπο. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. 2 Δεκεμβρίου θα συζητήσουμε το σχέδιο έκθεση του κυρίου Τάκουλα. Μετά τα υπόλοιπα τον Ιανουάριο. Λοιπόν, μετά το Δεκέμβριο δηλαδή θα έχουμε την επίσημη έκθεση του συναδελφού. Ευχαριστώ. Ως έμειναν, ξέρω πως είναι πέμπτη αργά. Απόψε έχω και το βραβείο λογοτεχνίας της Κομισιόν. Που θα πάω, πρέπει να είμαι αναγκασμένο να πάω και εκεί. Λοιπόν, 10 έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών, τα έχετε μπροστά σας, αν κανείς δεν έχει αντίρρηση εγκρίνονται 11 διάφορα δεν νομίζω να υπάρχει τίποτα στα διάφορα τελειώσαμε και με αυτό 12 ημερομηνία διαγωγής της επόμενης συνεδρίασης 1 Δεκεμβρίου 3 η ώρα 2 Δεκεμβρίου το πρωί τίποτα άλλο όχι ευχαριστώ ευχαριστώ και του διερμηνείς για το ότι έπρεπε να μεταφράσουν αυτές πολύ γρήγορε παρεμβάσει και υπέμειναν τα αγγλικά και τα γαλλικά μου σας ευχαριστώ, καλό ταξίδι στην περιφέρειά σας, καλές συναντήσεις να έχετε με τους ψηφοφόρους για σας.